Dear colleagues, please take your Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ήδη έχουμε 10 λεπτά καθυστέρηση. you. Thank you very much. I open the... Ωραία. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής μας και χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ σήμερα. Μετά στην ψηφοφορία φαντάζομαι ότι θα έρθουν και περισσότεροι. Αρχίζουμε λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. σχόλια. Όχι, εντάξει. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Πρακτικά της προηγούμενη συνεδρίασής μας, τη 13 η και 14 η Ιουλίου. Ως ήθιστε, αν δεν υπάρξουν ε, αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής, θα εγκριθούν. Τέταρτο σημείο. Είναι τεχνικής φύσεως, αλλά πολύ σημαντικό. Πρόκειται για την έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας για το 2016. Θα έχετε δει το σχέδιο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπονηθεί ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα για όλες τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Νομίζω ότι είναι καλύτερα το 2016 από ό,τι είχαμε για το 2015. Έχουμε λιγότερες πέμπτες να συνεδριάσουμε αλλά έτσι καλλιώς ήταν θέμα του Προεδρείου ε, φέτος για να για του χρόνου, γιατί τρίτη απόγευμα και τετάρτη πρωί δεν ήθελε συνεδρία στο Προεδρείο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο έχω παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι ότι ανακοινώσατε ότι θα είχαμε λιγότερε πέμπτε στην ημερήσια διάταξη, ενώ τώρα βλέπω ότι έχουμε πολλέ πέμπτε συνεδρίαση για την επόμενη χρονιά πως θα τα καλύτερα να το βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Είναι λιγότερες φέτος από ό,τι πέρυσι. Λίγο λιγότερες. Η κυρία Κρέλ. Ναι, ισχύει. Τρεις είναι οι πέμπτες με συνεδριάσεις επιτροπών. Ελέγξτε το κι εσείς, γιατί Συζήτησα και με ανθρώπους από άλλες επιτροπές και έχω πάλι την αίσθηση ότι είναι πάρα πολλές οι πέμπτες σε σύγκριση με τις άλλες επιτροπές. Και συγγνώμη, ε, μου είναι δύσκολο να το αποδεχτώ αυτό. Ίσως στην διάρκεια των επόμενων εβδομάδων ή μηνών θα μπορούσαμε κάποια από αυτές τις συνεδριάσεις πέμπτης να τις αλλάξουμε και άλλωστε κάποιες φορές ε, συμβαίνει να έχουμε λιγότερη δουλειά και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συμπτύξουμε κάποιες συνεδριάσεις τις άλλες μέρες ώστε να μην συνεδριάζουμε τόσο πολλές φορές την Πέμπτη. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να σας πω ότι θα γράψω στις αρμόδιες υπηρεσίες, αρμόδιες για το χρονοδιάγραμμα αυτό και θα τους πω ότι έχουμε πολύ σημαντικές δυσκολίες με τις συνεδριάσεις της Πέμπτης και να φροντίσουν να υπάρξει κάποια αλλαγή. Συμφωνείτε? Ωραία. Και θα σας στείλω φυσικά και το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής. Σημείο 5. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Τρεις ανακοινώσεις έχω να σας κάνω. Πρώτον, Η κυρία Μόνικα Σμόλκοβα δεν θα μπορεί να είναι εδώ από τους σοσιαλιστές, ζητά συγγνώμη. Δεύτερον, συνεδρίασαν οι συντονιστές σήμερα το πρωί πριν πάμε για την ψηφοφορία και τις αποφάσεις σα σας τις στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σήμερα ακόμα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Και η τρίτη πληροφορία που θέλω να σας δώσω είναι να σημειώσετε ότι στις 15 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο θα φιλοξενήσει μια τελετή για υπογραφή μιας ε, νέας συμφωνίας Covenant of Mayors. Θα γίνει στην αίθουσα της Ολομέλειας. Είναι μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τους στόχους, τους ενεργειακούς και τους κλιματικούς ε, σε τοπικό επίπεδο. Ήδη 6.000 ευρωπαϊκές πόλεις και δήμοι συμμετέχουν. Ένα αντίστοιχο γεγονός φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 2013. Ίσως κάποιοι από εσά να ήταν εκεί. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που είχα να σας κάνω. Δεν έχω άλλες. Προσπαθώ να πάω γρήγορα, διότι έχουμε εδώ έναν πολύ καλό φιλοξενούμενο σήμερα μαζί μας. Πρόκειται για τον Υπουργό για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Υποδομές και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε ακριβώς ε, μαζί του, ε, προεδρεύων ε, του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά και θα συζητήσουμε για την πολιτική συνοχής. Ε, μάλιστα συναντήθηκα μαζί του γιατί δέχτηκα πρόσκληση να πάω χτες και να μιλήσω σε διάσκεψη για τα 25 χρόνια του Ιντερέγκ. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί στο πρόγραμμα της Λουξεμβουργιανή Προεδρίας και πολύ θα ήθελα να ακούσω περισσότερα σήμερα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και εισαγωγή θα δώσω το λόγο στον Υπουργό. Ε, θα ακολουθήσει μετά την παρουσίασή του ε, συζήτηση. Μπορείτε να υποβάλλετε σχόλια και ερωτήσεις. Αλλά θα περιορίσω το χρόνο των παρεμβάσεων. Κύριε Ζηρά, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Με πολύ χαρά έρχομαι εδώ για να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητές μας και την πολιτική μας όσον αφορά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή. Θα αρχίσω πρώτα με την ε, συνοχή. Με τους φίλους μας από την Ιταλία και τη Λετωνία, από το 2013 και μετά έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα τριμερές στον τομέα της εδαφικής συνοχής. Επίσης ασχοληθήκαμε και με τις αστικές περιοχές. Είναι η πρώτη φορά. Αυτό το τρίο λοιπόν είχε μεγάλη ευθύνη γιατί έπρεπε να ολοκληρώσουμε τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει από συζητήσεις για το πώς μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Συνοχής, έτσι όπως συμπεριλαμβάνονται στις συνθήκε, για την εδαφική συνοχή. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η εφαρμογή πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και ετοιμαζόμαστε για την άτυπη συνάντηση με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μέσα για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της ε, συνοχής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία σε τρεις κυρίως τάσεις στον τομέα αυτών της εδαφικής συνοχής. Πρώτον, θέλουμε πρωτοβουλίες για σταδιακή σημασία συζήτηση όσον αφορά τα διάφορα σενάρια που μπορούν να υπάρχουν για την πρόοδο στην εδαφική συνοχή. Θέλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική συζήτηση που γίνεται όσον αφορά τα διάφορα σενάρια αυτά υπέρ της εδαφικής συνοχής ενώπιση του 2050. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την ανάπτυξη πολιτικών, όπως είναι η ενημέρωση της εδαφική ατζέντα για το 2020. Αναγνωρίστηκε όμω ο συγχρόνος ότι αυτή η εδαφική ε, διάσταση πρέπει να συνάδει με τις πολιτικές προτεραιότητες. Μία από τις κύριες αδυναμίες τη στρατηγική για την Ευρώπη το 2020 είναι ότι ακριβώ δεν αναγνωρίζει την εδαφική διάσταση. Η ανάπτυξη όμως εξαρτάται πολύ περισσότερο από τους περιφερειακούς παράγοντες. Πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς έτσι ώστε να εξοικειωθούμε περισσότερο με το θέμα. Έπειτα, η νομοθεσία για τις ε, για περιφερειακές περιοχές και διασυνοριακές περιοχές. Πρέπει να βελτιώσουμε συγχρόνως τι συνθήκε ζωής των πολιτών. Συνεπώς χρειάζεται μια νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση που να προσφέρει τα νομικά μέσα που θα δώσουν στι τοπικέ και περιφερειακέ αρχές τη δυνατότητα να προτείνουν στι χώρες μέλη λύσει για να αρθούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία. Πρέπει βέβαια να βασιστούμε στην υπάρχουσα νομοθεσία, στις προδιαγραφές που ισχύουν στις χώρες μέλη και να υπάρξει ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να εφαρμόζεται στα διάφορα προγράμματα τα διασυνοριακά. Πρέπει να συλλέξουμε παραδείγματα από τέτοια διασυνοριακή συνεργασία. Θα ανταμελετήσουμε λοιπόν και θα δούμε κατά πόσο είναι εφικτά αλλού και θα φροντίσουμε να εγκριθούν από τις ενδιαφερόμενες χώρες μέλη. Το πλαίσιο του EGCC είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ και πρέπει να ξέρουμε ότι δεν το αντικαθιστούμε εμείς. Δρούμε συμπληρωματικά. Τώρα για το ρόλο των ε, μικρών και μεσαίων πόλεων υπέρ της ανάπτυξης της Ευρώπης. Ο ρόλος τους αγνοείται σε ένα μεγάλο βαθμό στον πολιτικό λόγο μέχρι σήμερα, παρόλο που οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Η Λουξεβοριανή Προεδρία ε, το ξέρει, γιατί ξέρει πόσο πολυκεντρικό δίκτυο είναι το Λουξεμβούργο και πώς μπορούν οι μικρές και μισές πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους. Είναι κάτι που δείχνει επίσης ότι η εδαφική και η αστική πολιτική συνδέονται μεταξύ τους. Από πλευράς πολιτικών λοιπόν, το βασικό είναι η αστική ατζέντα. Πώς την αστική διάσταση θα τη υπόψη μας στις πολιτικές μας, ώστε οι πολίτες που ζουν στις πόλεις να μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους, ώστε να επιτεθούν οι στόχοι της Ευρώπης το 2020. Η αστική ατζέντα θα εντοπίσει λοιπόν τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και θα δούμε ποιες από αυτές έχουν τη μεγαλύτερη προσπιθέμενη αξία. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την επερχόμενη Ολλανδική Προεδρία επί του θέματος. Η μεγαλύτερη πόλη στο Λουξεμβούργο έχει 100.000 πολίτες, οπότε ίσως ε, η Ολλανδική Προεδρία να δει αλλιώς τις μεγάλες πόλεις Γι' αυτό πάντως τους αφήνουμε και τη δυνατότητα να οργανώσουν μεγάλες εκδηλώσεις την άνοιξη που μας έρχεται. Υπάρχει και έκθεση του Κοινοβουλίου που δεν την έχουμε αξιολογήσει πλήρως ακόμα. Όταν ε, πάντως εξετάζουμε το θέμα της αστικής ατζέντα, τις μικρές και τις μεγάλες ε, πόλεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την Ήπεθρο, γιατί και εκεί υπάρχουν ε, χώροι για τους πολίτες μας και πρέπει να έχουμε υπόψη μας θέματα όπως είναι η ενεργειακή αποκέντρωση. Για το Ιντερεκ τώρα πιο συγκεκριμένα θέλω να επενθυμίσω την μεγάλη εκδήλωση αυτή της Προεδρίας τις τελευταίες δύο μέρες την οποία ήρθε και η Πρόεδρος. Γιορτάσαμε τα 25 χρόνια λοιπόν του Ιντερεκ. Πάνω από 500 άνθρωποι ήρθαν από τις 28 χώρες μέλη. Ήτανε και για να γιορτάσουμε αλλά και για να προβληματιστούμε προκειμένου να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματα του Ιντερεκ, πώς, έχουν, πώς έχει αλλάξει η πολιτική από τότε που ξεκίνησε το 1990 ως κοινοτική πρωτοβουλία και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Και πολύ χαρήκαμε που σας είχαμε μαζί σας κύριε Πρόεδρε. Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα εξεταστούν τον Νοέμβριο στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα τις μακροπεριφερειακές πρωτοβουλίες, εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ε, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τα συμπεράσματα για τις περιφέρειες των Άλπων. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ικανοποιητικά τη στρατηγική μας με ένα καλό συντονισμό ε, στην Ευρώπη και με άλλα επενδυτικά ταμεία. Θα στραφώ τώρα στην πολιτική συνοχή. Το Λουξεμβούργο βέβαια είναι μια ε, μικρή χώρα, δεν είναι μεγάλη σημασία όμως στα διευθυντικά ταμεία. Παρόλο που το ίδιο το Λουξεμβούργο δεν τα χρησιμοποιεί πολλά. Πιστεύουμε ότι αποτελούν μια προστεθέμενη αξία πολύ σημαντική για την ε, ανάπτυξή μας και για τους στόχους του 2020. Και είναι σημαντικό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι προτεραιότητές του μέχρι το 2020. Εδώ έχουμε υπόψη μας και το ευρωπαϊκό εξάμεινο προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σημειώνουμε επίσης την πρόοδο αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη. Ως Προεδρία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την πολιτική συνοχή και θα συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων προεδρίων και θα ολοκληρώσουμε με το νομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Παραμένουν ε, κατεξουδότηση πράξης βέβαια στο πακέτο των διαθετικών ταμείων. Η Προεδρία επίσης θέλει λύσεις για ειδικά μέτρα στην πολιτική συνοχή και μπορώ να σας ανακοινώσω με χαρά σήμερα ότι το Συμβούλιο πρόσφατα αποφάσισε να επιταχύνει την έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις διατάξεις για την Ελλάδα. Πρόκειται για έκτακτα μέτρα και πρόκειται βέβαια για μια μοναδική κατάσταση η οποία οφείλεται στην ε, κρίση και γι' αυτό είναι σημαντικό από τα διορθωτικά ταμεία, τα επενδυτικά ταμεία να υπάρχουν αρκετά ποσά τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν πραγματικά για επενδύσει επιτόπου, ώστε να αποφεληθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι πολίτε εκεί. Ξέρω ότι και εσεί είσαστε υπέρ του ίδιου στόχου. Γι' αυτό θέλω να αποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να σα ευχαριστήσω όλου για την καρποφόρα συνεργασία η οποία οδήγησε σε αυτήν την γρήγορη θεσμική συμφωνία και σε γρήγορη εφαρμογή. Θα ξέρετε ίσως ότι χτες στην Κορεπέρ βρήκαμε λύση για αυτά τα ζητήματα. Έρχομαι τώρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Βασιστήκαμε στα επιτεύγματα της Ιταλικής Προεδρίας και είχαμε το πρώτο Συμβούλιο πέρυσι για την πολιτική συνοχής. Εμείς θέλουμε να συνεχιστούν δομημένες συζητήσεις στο Συμβούλιο όσον αφορά τη συνοχή και όχι μόνο κάθε φορά που συζητούνται νέες ρυθμίσεις, νέοι κανονισμοί. Θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνεισφορά των διεθντικών και επενδυτικών ταμείων υπέρ της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές και ως Λουξεμβουριανή Προεδρία θέλουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής να ληφθεί υπόψη παντού. Ίσως θα τα ακούσατε και από το ΕΚΟΦΗΝ και στο Συμβούλιο Γεωργίας, γιατί βέβαια η κλιματική πολιτική δεν είναι θέμα μόνο των Υπουργών Περιβάλλοντος. Πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις πολιτικές. Η πολιτική συνοχής επίσης θα είναι κεντρικό θέμα όσον αφορά την επίτευξη των κλιματικών μας προτεραιοτήτων. Συνεισφέρουμε λοιπόν στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του COP21 που θα λάβει χώρα στο Παρίσι στα τέλη της χρονιάς. Κάτι άλλο για το Σεβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η προσθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας. Αυτό είναι το Ίντερεγκ βασικά. Ποιο θα είναι το μέλλον του Ίντερεγκ λοιπόν ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία του. Και εδώ φτάνουμε στα συμπεράσματα που ανέφερε αρχικά και η Πρόεδρος, τα συμπεράσματα της διάσκεψης που είχαμε στο Λουξεμβούργο χθες και προχθές για 25 χρόνια Interreg. Πιστεύουμε ότι το Interreg θα έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον για να πετύχει την συνέχεια, τη συνοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο για το Γενικό Συμβούλιο είναι η συζήτηση πιο περίπλοκων θεμάτων όπου εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φτιάξει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου προκειμένου να παρουσιάσουν τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των χωρών μελών. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα έχουμε αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές, ο κ. Βανίστερλόι. Έχουμε τη δυνατότητα να... να σας επαναλάβω ότι πρέπει να είστε λακωνικός. Ναι, βεβαίως. Σα ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και να κάνω κάποια σχόλια. Μιλήσατε για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Είναι σημαντικό τα συμπεράσματα της ρήγα να γίνουν απόλυτα και άμεσα ε, αποδεκτά, Ούτω ώστε να έχετε τα συμπεράσματα. Ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα της Ιταλικής Προεδρίας. Επίσης, δεν έχετε άτυπη συνάντηση των Υπουργών για τη συνοχή αυτή την περίοδο. Θα πρέπει δηλαδή να κάνετε αμέσω τη συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Για ποιο λόγο. Μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια να το σχολιάσετε. Μία παρατήρηση τώρα για την εδαφική διάσταση και τη συζήτηση που γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κρίμα που λείπει την έκτη έκθεση για τη συνοχή της Κομισιόν. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε εσείς και οι συνάδελφοί μου νομίζω θα επανέλθουν στο θέμα αυτό. Η εδαφική συνεργασία θα είναι ακόμα πιο σημαντική στο μέλλον. Σε πράγματα που δεν μπορούμε να ε, φανταστούμε τώρα, γιατί είναι κλασικά ευρωπαϊκά θέματα αυτά και αφορούν τους πολίτες μας. Τους μας. Τρίτη παρατηρήση. Δεν μίλησα για το ΕΦΣΥ. Θα κάνει κάτι το Λουξεμβούργο. Ψάχνετε τους ανθρώπους ε, που θα έρθουν ε, για να υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτως ώστε να γίνει κάτι σημαντικό. Είναι κάτι που θα πρέπει να κάνει το Λουξεμβούργο. Το βασικό μας όμως θέμα, και το έχουμε συζητήσει και αλλού, σε άλλες συνεδριάσεις, είναι οι συνέργειες ανάμεσα στο νέο ταμείο, ε, το οποίο συνδέεται με το ένα και το άλλο, με, με το ένα και το άλλο ταμείο εννοώ, με διάσπαρτο τρόπο. Πώς δημιουργούνται οι συνέργειες οι απαραίτητες. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για τα, τους τρεις άξονες που αναφέρατε κύριε Φυπουργέ και είπατε ότι θέλετε να επεξεργαστείτε στην διάρκεια της προεδρής σας. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι Ακολουθείτε με μια κάποια καθυστέρηση της ε, προτεραιότητας του Κοινοβουλίου γιατί το προηγούμενο διάστημα εμείς είχαμε ε, επισημάνει αυτούς ακριβώς τους ε, άξονες ως τους σημαντικούς. Εν πάση περιπτώσει σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Λοιπόν, για την συζήτηση, τη στρατηγική συζήτηση για την εδαφική συνοχή. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι ακριβώς σας ενδιαφέρει οικονομικά στοιχεία, πληθυσμιακά. Δεύτερον, αν κατάλαβα σωστά, θέλετε τροποποίηση του κανονισμού για τη διασυνορική συνεργασία. Το χαιρετίζω αυτό. Αλλά, αν θέλετε να προβλέψετε νέες υποδομές, να φροντίσετε και τα χρήματα να υπάρχουν. Ε, γιατί εμείς στις διαπραγμα... διαπραγματεύσεις, το είχαμε ζητήσει αυτό χωρίς την υποστήριξη του Συμβουλίου στις διαπραγματεύσεις, Όσον αφορά την, ε, ε, την αστική ανάπτυξη και το σχετικό ψήφισμα που εγκρίναμε, ε, θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλλει στην γενικότερη συζήτηση. Και αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω είναι την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο να λάβει απόφαση επιτέλους για τους πρόσφυγες που είτε έχουν έρθει είτε θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και θα ήθελα να σας ζητήσω να υπάρξει μια πρωτοβουλία ώστε τα κράτη-μέλη να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούν ε, κονδύλια ευρωπαϊκά το επόμενο διάστημα με ευελιξία πάντοτε προκειμένου να υποδεχθούν, να εγκαταστήσουν, να ε, εκπαιδεύσουν τους πρόσφυγες, να τους παράσχουν υγειονομική περίθαλψη και να μην ε, εξαφανιστείτε τις επόμενες... Ε, οι, οι πρόσφυγες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν τις επόμενες εβδομάδες. Θα είναι μαζί μας για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι χρειάζεται μια ευελιξία στο πώς τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αξιοποιούν τα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Τόμασιτς. samo zanima jedno najviše sada Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση που είναι η πιο σημαντική για μένα. Χθε ε, στην Κροατία ξαφνικά αρχίσαμε να λαμβάνουμε πρόσφυγες. Χιλιάδες. Περιμένουμε ότι θα έρθουν 10 με 100 χιλιάδες. Και για μια χώρα όπως η Κροατία που έχει 4 εκατομμύρια ε, κατοίκους θα ήταν καταστροφή κάτι τέτοιο. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα και πώς θα βοηθήσετε τις ε, πιο φτωχές χώρες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Ποιος uh, Βαν Καλώς ορίζουμε τη Λουξεμβουργιάτικη Προεδρία, φυσικά. Σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις σας. Τα τρία σημεία που αναφέρατε, που μπορεί να συμπεριληφθούν σε συμπεράσματα του Συμβουλίου, είναι πολύ πολύτιμα. Σας ευχαριστώ που δίνετε σημασία στην κλιματική προσαρμογή και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για μια χρήσιμη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθωτικών και επενδυτικών ταμείων που να έχει και επιπτώσεις. Αν χάσουμε έξι μήνες επί Λουξεμβουργιάζικης Προεδρίας και περιμένουμε την επόμενη Προεδρία, την Ολλανδική, να συνεχίσει το follow-up της δήλωσης της Ρήγας, θα ήταν κρίμα πραγματικά. Θα έλεγα λοιπόν να προετοιμαστείτε μαζί με την Ολλανδική Προεδρία ε, για μια ατζέντα εφαρμογής, ούτως ώστε να αρχίσουμε από τις αρχές του 16 με τη Ρήγα. Ε, Έχουμε επίσης μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά την πολιτική, ε, την εργατική, σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ για να ενισχύσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ειδικά σε μεθοριακές περιοχές. Τελευταίο σημείο. Η απλούστευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι είναι αρκετά χρήσιμο να μιλάμε όχι μόνο σε ομάδα υψηλού επίπεδου, αλλά και με του συναδέλφου σας, ε, για την απλούστευση της διαχείρισης των ταμείων και να δώσουμε μία πνοή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το περιμένουν από μας. Γιατί το τελευταίο που θέλουμε στην Ευρώπη είναι να διώξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην χρησιμοποιούν τα διαφθορτικά ταμεία. Ε, κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι για τη συζήτηση που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή. Ένα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την Επιτροπή μας το να γίνει ένα άτυπο Συμβούλιο που να ασχοληθεί με την ε, συνοχή δείχνει την σημασία και την προτεραιότητα που δίνεται στην πολιτική αυτή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια από τις σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε κι εσείς ότι το Λουξεμβούργο είναι μια χώρα που δεν καταναλώνει ουσιαστικά τα διαστοτικά ταμεία. Ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε με, μεγάλη, με μεγάλο ενδιαφέρον τη δέσμευσή σας για τα θέματα αυτά. Μιλήσατε για πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω και από το πιο σημαντικό ερώτημα για την Ευρώπη. Αλλά και για τις περιφέρειες της Ευρώπης, που είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Δεκέμβριο θα γίνει η διάσκεψη του Παρισιού. Ξέρουμε σήμερα ότι αν ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε τρομερά προβλήματα που θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Και η αύξηση του επίπεδου των ωκεανών μπορεί να ξεπεράσει το ένα μέτρο. Μερικοί εμπειρογνώμονες μιλούν για τέσσερα ή πέντε μέτρα η περιφερειακή πολιτική μπορεί να αποσταθεροποιηθεί όταν ξέρουμε ότι το σύνολο ή τουλάχιστον πάρα πολλές υποδομές, ε, ανάπτυξη βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία είναι πολύ εκτεθειμένη στο νερό. Βρέχεται από πολλές πλευρές ε, από θάλασσες και ωκεανούς. Τι θα κάνετε ούτως ώστε να εφαρμόσετε μια πραγματική στρατηγική ευρωπαϊκής ε, διάστασης, περιφερειακή στρατηγική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, το είπατε και εσείς, κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Είναι το θέμα των μεταναστών φυσικά και των προσφύγων που έρχονται και αποσταθεροποιούν κάποια στοιχεία της ε, περιφερειακής πολιτικής. Βλέπουμε ότι η περιφερειακή πολιτική επιτρέπει να μετριάσουμε κάποιες επιπτώσεις και να, δώσουν, να δώσει και κάποιες λύσεις. Παραδείγματο χάρη στην Ιταλία. Το Συμβούλιο θα υποστηρίξει την Κομισιόν στον προβληματισμό που έχει ξεκινήσει ήδη σήμερα, ούτω ώστε οι πιστώσεις ε, της συνοχής να μπορέσουν να εισρεύσουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα προτεραιότητα, που είναι πάνω απ' όλα η υποδοχή των προσφύγων. Τελευταίο σημείο, το είπατε επίσης, αφορά την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ αντιδραστικό, συγγνώμη, ε, και το Κοινοβούλιο και για το θέμα της Ελλάδας και το θέμα των προσφύγων. Η πολιτική συνοχής είναι αυτή η οποία μπορεί να λειτουργήσει και να μετριάσει κάποιες βίες επιπτώσεις ε, ευρωπαϊκών πολιτικών, άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Βασιστείτε πάνω μας, εάν θελήσετε να προτείνετε τέτοιες λύσεις έτσι, πραγματικά θετικές. Ευχαριστώ κύριε Βάνα. Ευχαριστώ Καλώς ήρθατε κύριε Φιβουργέ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για, τις, ε, για την παρουσία σας. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Λουξεμβουργιανή Προεδρία υιοθετεί μια προσέγγιση στρατηγικού χαρακτήρα για την πολιτική συνοχής, διότι πράγματι δεν μιλούμε μόνο για την τεχνική εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και για την ε, εδαφική, ε, οικονομική και κοινωνική συνοχή της ε, Ευρώπης. Αυτή είναι άλλωστε η ουσία της πολιτικής συνοχής, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης, όπου σε κάποιες χώρες ε, τα μια αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων επενδύσεων. Άρα χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Μιλήσατε και για την κλιματική αλλαγή και οι προλαλήσαντες ε, σας έθεσαν κάποια θέματα σχετικά. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Στο πρόγραμμα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας ε, γίνεται αναφορά στο Greening the European Semester, πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, που βεβαίως θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ως στόχος. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα πάρετε αφενός και αφετέρου ε, θέλω να μου πείτε τις ε, προθέσεις σας σε σχέση με τις μεθοριακές περιοχές. Είπατε κάτι και για έναν καινούριο κανονισμό. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα να μας πείτε. Και δεύτερον, ε, αν μπορείτε να μας πείτε ε, τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλυθούν για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων ε, πόλεων. Ε, επίσης είδα ότι στο πρόγραμμα της Προεδρίας ε, ε, υπάρχει η πρόθεση να ενισχυθεί και η έρευνα στον τομέα του gender mainstreaming. Και εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Πείτε μας κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Δεν θα επαναλάβω ερωτήματα τα οποία έκαναν συναδελφοί μου και που με κάλυψαν. Ένα πράγμα μια και μεταξύ των προτεραιοτήτων του Λουξεμβούργου είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων και άρα να υπάρξει ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα να, σας ρωτήσω πώς θα εφαρμόσετε το, περί, το περίφημο σχέδιο ΕΦΣΙ για τα διαβόητα 315 δις. Πέρα από τη γνώση της, ε, γνώμη της Κομισιόν που την ξέρουμε, ποια είναι η άποψη των 100 μελών και τι, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα αυτό, έτσι, των 315 δις και τι ευραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μπορούμε να περιμένουμε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Ναι, γνωρίζω. Απλά θέλω να τελειώσουμε πρώτα με τις ερωτήσεις των συντονιστών. Άρα, ολοκληρώθηκε αυτός ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στον προσκεκλημένο μας και στη συνέχεια θα μπορέσετε να θέσετε τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Δεν είχαμε χρόνο να διοργανώσουμε άτυπη συνάντηση για την πολιτική συνοχή. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ε, ημερομηνία ακόμα και για, την, ε, για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αν δείτε, ε, ε, ε, όσε χώρε αναλαμβάνουν την Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο έχουν δύο μήνε λιγότερο και δυστυχώ ζητώ συγγνώμη αλλά δεν είχαμε τον χρόνο να διοργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση. Ο κ. Μίσλ Ρόι υποστηρίζει και χαίρομαι γι' αυτό την ιδέα μα να υιοθετήσουμε μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική για την εδαφική συνεργασία και να προσπαθήσουμε να βρούμε και σε ποιους άλλους τομείς ε, η εδαφική πολιτική και η εδαφική συνοχή ε, έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι που δεν ε, έχει γίνει στο παρελθόν και εμείς τουλάχιστον ως Προεδρία θα το προσπαθήσουμε. Στο Λουξεμβούργο υπάρχουν πάρα πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Το έξι βεβαίως θα έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο ε, και αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξουν συνέργειες ε, προκειμένου να επιτεθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Θέλουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να υπερβούμε τυχόν εμπόδια που θα εμφανιστούν στο δρόμο μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές οι ε, συνέργειες. Για την κυρία Κρυλ καταρχάς να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζεται αυτούς τους τρεις άξονες που παρουσίασα. Εχθές στο σεμινάριο του Ίντερεγ μας ε, υπόθηκε ότι αναφέρθηκε ότι πολλές φορές στην αρχή ε, το Interreg θεωρούνταν από πολλούς ως ε, μια χρυσή αγελάδα την οποία μπορούσαν να αρμέγουν. Μια αγελάδα που βρισκόταν εδώ στις Βρυξέλλες για να παίρνουν λεφτά. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Και όπως είπατε και εσείς, όταν κανείς υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη ε, στρατηγική επενδύσεων θα πρέπει να έχει και ένα όραμα για το που θέλει να πάει. Και αυτό είναι προφανές ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τα πάνω. Γιατί αν θέλουμε να οραματιστούμε, ε, αν θέλουμε μάλλον, πρέπει μάλλον να έχουμε ε, ένα όραμα για την Ευρώπη, για το πώς θέλουμε να είναι σε 20 και 30 χρόνια, προκειμένου αυτή να μπορέσει στη συνέχεια να εξειδικευθεί και σε εδαφικό επίπεδο. Γιατί ε, χρειαζόμαστε ε, ένα τέτοιο όραμα λοιπόν. Ξέρετε ότι ξεκίνησε λοιπόν αυτό το έργο στο Λουξεμβούργο για να ξεκινήσει ε, αυτή η ανάπτυξη ε, της πολιτικής συνοχής, της ε, εδαφικής συνοχής και έχουν, αναφερθεί, έχουν αναλυθεί τρία σενάρια. Πρώτο σενάριο, ε, ανάπτυξη μόνο των Μητροπόλεων, ανάπτυξη της υπαίθρου και ανάπτυξη των ε, λιγότερο ανεπτυγμένων ε, περιφερειών. Αυτά είναι τρία διαφορετικά σενάρια. Το ποιο σενάριο θα επιλέξουμε από στρατηγικής άποψης θα έχει ε, επιπτώσεις στο πώς θα δαπανηθούν, πώς θα επενδυθούν τα χρήματα στους διάφορους τομείς πολιτικής. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν, ιδιαίτερα ε, με βάση το κεκτημένο που υπάρχει μπορούμε να βασιστούμε στο έργο που έχει προηγηθεί στο παρελθόν, στο πλαίσιο του ίντερνετ και νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα κάνουμε εμείς. Πολλοί ρώτησαν πώς φανταζόμαστε αυτό το πρόσθετο εργαλείο για την ε, διεθνική συνεργασία. Είχα πάει και στην Επιτροπή των Περιφερειών ε, πρόσφατα και είδα ότι υπήρξαν και εκεί πολλές επιφυλάξεις. Γνωρίζουμε δύο πράγματα πρέπει να σας πω. Πρώτον, αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μια νυχτή. Είναι ένα, μια ιδέα μέσω μακροπρόθεσμης ε, υλοποίησης και χρειαζόμαστε βεβαίως διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες γιατί πολλά ζητήματα έχουν παρερμηνευτεί. Πρώτον, δεν πρόκειται για εργαλείο που δρά ανταγωνιστικά προς το ETGC. Είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα που το έχετε ζήσει κι εσείς. Ε, εγώ ήμουν ε, 20 χρόνια δήμαρχος σε μια μικρή πόλη. Κάποια στιγμή λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα ε, να ε, πάρουμε τα ε, ε, λίματα ενός μικρού βελγικού χωριού που βρισκόταν πολύ κοντά μας και τα οποία μπορούσαμε να ε, επεξεργαστούμε εμείς στις δικές μας ε, εγκαταστάσεις. Όταν έμαθα ότι χρειαζόμαστε διακρατική συμφωνία για να γίνει κάτι τέτοιο, να φέρνουμε τα λίματα από ένα μικρό βελγικό χωριό στη δική μας πόλη που ήταν πάρα πολύ κοντά, φυσικά δεν συνέχισα. Άρα, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Φανταστείτε το. Το βελγικό αυτό χωριό θα έπρεπε να αιτηθεί στις δικές της ε, αρχές ε, για έγκριση, να αιτηθεί έγκριση και το Λουξεμβούργο στις δικές του αρχές. Πάντως, αν οι διαδικασίες αυτές μπορούσαν να επιταχυνθούν, θα μπορούσαν ένα τέτοιο έργο να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερες συνεργασίες, ιδιαίτερα στι περιοχές, περιοχέ, μεθοριακές περιοχές ε, περιοχές. Αλλά η συζήτηση θα πρέπει να φύγει από αυτό το αφηρημένο επίπεδο και να δούμε τι ακριβώς επιπτώσεις θετικές μπορεί αυτή η συνεργασία να αποφέρει στους ίδιους τους πολίτες. Τρίτον και θα ήθελα να τοποθετηθώ με αυτό ε, για την ε, κρίση με τους πρόσφυγες. Προφανώς δεν είναι ούτε η ώρα ούτε ο τόπος εδώ να ε, επιλύσουμε το πρόβλημα οριστικά. Αυτό που θέλω όμως ε, είναι να σας ζητήσω να είστε σύμμαχοί μας στο Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με ευελιξία τα ταμεία ε, και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε οι χώρες δηλαδή που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές να μπορέσουν να έχουν μια ε, ευελιξία στην αξιοποίηση των κονδυλίων. Για τον κύριο Μίλτινμπαρκ. από τις κάτω χώρες. Νομίζω ότι ε, με παρερμηνεύσετε όσον αφορά την αστική ατζέντα. Δεν είπα ότι δεν θα εργαστούμε τους έξι μήνες αυτούς στην, ε, στον τομέα της αστικής ατζέντα. Αντιθέτως, οι Ολλανδοί συνάδελφοί μας έχουν αναλάβει ηγετική πρωτοπόρα θέση, έχουν μεγάλη εμπειρία. Σε συνεργασία λοιπόν με τους Ολλανδούς φίλους μας, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τους επόμενους έξι μήνες αυτήν την αστική ε, ατζέντα. Για την ε, αγορά εργασίας. Είχαμε κάποια πολύ καλά παραδείγματα ε, τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα σε Πολωνία και Γερμανία το πώς μπορούν να, μέσω του Ίντερεγ να δημιουργηθούν κοινέ αγορές εργασίας και το Λουξεμβούργο είναι επίσης μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό παράδειγμα και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δείξουμε πώς ε, καθημερινά υποδεχόμαστε 170.000 εργαζόμενους από τις τρεις γειτονικές μας χώρες. Ε, αυτό βεβαίως δημιουργεί και μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Λουξεμβούργου, αλλά είναι και, μια μεγάλη, είναι και ένα μεγάλο επίτευγμα, γιατί πρόκειται ε, από γεωγραφικής άποψης για το μεγαλύτερο χώρο ε, μετακίνησης εργαζομένων, άρα το κατανοούμε πλήρως την προστιθέμενη αξία μιας πολιτικής για την ε, μεθοριακή συνεργασία. Ε, όταν ήμουν δήμαρχος ε, σε αυτήν τη μικρή πόλη πρέπει να σας πω ότι ε, αντιμετώπισα στην πράξη πόσο δύσκολο είναι να γίνεται μια διαχείριση όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις μικρές πόλεις το, πώς, ε, το να συμμετέχει κανείς σε ευρωπαϊκά έργα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ε, έργα να έχουν τη δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του κυρίου Μαζέ, κατάλαβα ότι για μας ε, η κλιματική αλλαγή είναι η Λουξεμβουργιαζική Προεδρία να ασχοληθεί όχι μόνο με την πολιτική συνοχή, αλλά να τα δει όλα αυτά μέσα σε ένα ολικό πλαίσιο, ολιστικό πλαίσιο. Και θα είναι και φταίξιμο της Ευρώπης αν δεν βρεθεί συνεργασία. Ε, η Γαλλική Προεδρία, ε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ε, πήγε μέσα σε μια μέρα να δει τον κύριο Φαμπιούς ε, και γύρισε την ίδια αυθημερών. Θα κάνουμε, για να δείτε δηλαδή πόση συνεργασία υπάρχει, ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να μην είναι η Ευρώπη αυτή που θα φρενάρει τις ε, διαπραγματεύσεις. Ο υπουργό έκανε πολλές διμερείς με διάφορες τρίτε χώρες. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές απροθυμίες, πολλοί δισταγμοί. Αυτό που θα κάνουμε πέρα από τις γενικές διαπραγματεύσεις είναι θα προσπαθήσουμε άπαξ και διαπαντός στη συμφωνία να μιλήσουμε για το σημαντικότατο ρόλο των περιφερειών και των κοινοτήτων. Συμφωνούμε απόλυτα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια συνολική δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι. Ε, αυτό είναι το πλαίσιο όμως. Ε, αύριο θα πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική μετριασμού και η πολιτική προσαρμογής. Και ποιος θα τις εφαρμόσει τις πολιτικές, οι πόλεις και οι κοινότητες. Οι δήμοι και οι κοινότητες. Ε, και χαίρομαι που η Προεδρία ανέφερε το σύμφωνο των ε, δημάρχων. Για μένα ήταν θαυμάσιο που είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε ότι για την πολιτική κλιματικής αλλαγής πρέπει να εμπλέξουμε τους Δήμους και τις κοινότητες της πόλης. Και εγώ ήρθα σε επαφή με τον κόσμο, με, τα, με τους υπαλλήλους ε, της Κομισιόν για να διευρύνουμε αυτό το σύμφωνο των δημάρχων και να κάνουμε ένα γενικότερο σύμφωνο, ούτως ώστε ε, και οι κοινότητες της ε, Νότιας Αμερική, Αμερικής, δηλαδή της Αμερικής και της Αφρικής να συνεργαστούν. Φανταστείτε ας πούμε τις διδημοποίησεις, φανταστείτε τις συνεργασίες που μπορούν να προκύψουν από κάτι τέτοιο. Μετά από τη συμφωνία που θα βρούμε, ελπίζω να βρούμε, ελπίζω να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα περισσότερε προσπάθειε, ούτω ώστε οι πόλεις και οι κοινότητες να έχουν πολύ περισσότερα μέσα, ούτω ώστε να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία. Για τους μετανάστες, προφανώ το Ταμείο Συνοχής μπορεί να βοηθήσει. Αλλά δεν θα το λύσουμε εδώ το πρόβλημα. Περιμένουμε την συνεισφορά τη Συνόδου Κορυφή, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Για την Ελλάδα συμφωνούμε. Χθε σα είπα ότι υπήρξε μια συμφωνία στο Κορεπέρ. Τώρα θα πρέπει να δούμε τα θεσμικά προβλήματα που υπάρχουν και η Κομισιόν θα πρέπει να τα επιλύσει. Φαντάζομαι ότι και εσείς και εμείς κάναμε πάντως μια καλή προσπάθεια. Ähm, äh, σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Ε, εν μέρη έχω απαντήσει. Το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την οικολογική επίπτωση άλλων θεμάτων. Δηλαδή, ε, κοινωνική συνοχή, οικονομικά θέματα, ανεργία. Όλα έχουν επιπτώσεις. Καλύτερα να αποφύγουμε την περιβαλλοντική ζημιά παρά να προσπαθούμε να την ε, διορθώσουμε μετά, να την παλώσουμε μετά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον τρίτο πυλώνα βιωσιμότητας που αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Σύνος Κορυφής της Νέας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης μας έδωσε καλούς δείκτες που θα πρέπει να εγκριθούν. Το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τους 17 στόχους βιωσιμότητας. Ε, και να μην αφορούν ε, μόνο τις χώρες του Νότου, αλλά όλες τις χώρες. Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους 17 στόχους βιωσιμότητας. Νομίζω Η πρώτη απόπειρα έγινε από κάτω, να φτιάξουμε το βάθρο για να ορίσουμε πιο συγκεκριμένα, ή μάλλον θα πρέπει να γίνει, για να δούμε τι σημαίνουν για μας αυτοί οι 17 στόχοι. Εμείς είμαστε μεταξύ ημών υπάρχουν πολλές χώρες, ή μάλλον στην κατάταξη του ΩΣΑ είμαστε στο μέσον κοιτάζουμε τους στόχους ε, της ε, βιωσιμότητας και θα πρέπει να δούμε πώς τους εφαρμόσουμε. Δεν κατάλαβα την τελευταία ερώτηση του, κυρίου, του κυρίου Αμάτο, της κυρίας Αμάτο. Ευχαριστώ. Ρωτούσα. Πώς η Προεδρία σας προτίθεται να εφαρμόσει το διαβόητο σχέδιο ΕΦΣΥ για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα αποτελέσματα, όχι. Τι μία απάντηση λέει ο Πρόεδρος. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω 7 συναδέρφους ακόμα στον κατάλογο μιλητών. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, όπως πάντα. Γι' αυτό σας παρακαλώ ένα λεπτό για την κάθε ερώτηση για να μας απαντήσει και ο υπουργό. Η κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω στο στο GST. Είναι μια δομή που πρέπει να περάσει από τις χώρες. Είναι ένας κανονισμός που πρέπει να εγκριθεί. Άμα εγκριθεί ο κανονισμός, γιατί να πρέπει επιπλέον να περάσει από τις χώρες μέλη. Αν θα μπορούσα να σας δώσω μια συμβουλή, θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να το καταργήσουμε. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη, είμαστε μια κοινή δομή, κοινέ οδηγίες, κανονισμούς. Οπότε δεν ξέρω τι προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει έγκριση από τις χώρες μέλη. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και μια τελευταία ερώτηση. Δεδομένου ότι θα εγκρίνεται την ε, μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις, η κλιματική προσαρμογή είναι πολύ σημαντικό. Συνδέεται. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να προσθεθεί και αυτή η διάσταση γιατί ξέρετε ότι οι ορεινές περιφέρειες είναι πάρα πολύ ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές. Άρημον, επόμενος ο μιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ έρχομαι από το Ανατολικό Βέλγιο, πολύ κοντά δηλαδή στο Λουξεμβούργο. Στην καθημερινότητά μου ως Ευρωβουλευτής έρχομαι αντιμέτωπος με υποθέσεις ανθρώπων που καθημερινά ε, φεύγουν από το Βέλιο και πηγαίνουν να δουλέψουν στο Λουξεμβούργο. Θέλω λοιπόν να δω κατά πόσο λειτουργεί πραγματικά η εσωτερική αγορά. Κάποιος που δουλεύει πάνω στις υποθέσεις των ανθρώπων αυτών θέλει να ξέρει γιατί δεν προχωράμε. Υπάρχει διαφορά στην νομοθεσία και δεν υπάρχει πάντα βούληση από τους πολιτικούς να αλλάξουν την νομοθεσία που είναι διαφορετική από τις δύο πλευρές των συνόρων. Τι έχει γίνει από αυτού. Πραγματικά δεν μπόρεσα να μάθω. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις. Εσείς τι σκοπεύετε τελικά να τροποποιήσετε ακριβώς για τέτοια προγράμματα όπως είναι το Interreg. Είναι αναγκαίο να γίνει η αλλαγή για να μπορέσει να επιβιώσει. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις ε, προτεραιότητές σας. Συμφωνώ με τόσα είπατε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην πολυκεντρική ανάπτυξη. Πρέπει να αναπτύξουμε και τις πόλεις και την Ήπεθρο. Αυτό είναι το κλειδί για τη σταθερότητα των διαφόρων χωρών. Εγώ είμαι από την ε, Σλοβενία και πάνω από το 50% των κατοίκων ζουν στην Ήπεθρο. Έχουμε υποδομές, αυτό που δεν έχουμε είναι δουλειές στην Ήπεθρο. Τα λέω όλα αυτά σε σχέση με την μετανάστευση και τους μετανάστες που έρχονται στην ε, Ευρώπη. Όμως μετανάστευση έχουμε και μέσα στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάνε σε μια άλλη. Άρα υπάρχει μετανάστευση και ενδοευρωπαϊκή, αλλά και μέσα και στην κάθε χώρα χωριστά. Συνεπώς, αν δεν υπάρξουν οι ίδιες συνθήκες για όλους, τόσο στις πόλεις όσο και στην Ήπεθρο, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Επιπλέον, πρέπει να επικεντρωθούμε και στις χώρες εκείνες οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Δυτικά Βαλκάνια δηλαδή. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, να βοηθάμε αυτές τις χώρες για να υπάρχει περισσότερη συνοχή και σταθερότητα. Ευχαριστούμε η κυρία Μισελ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, έχετε θέσει ένα πολύ φιλόδοξο στόχο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε αναγνωρίσει ως ε, σημαντικό τομέα την συμμετοχή των ε, τοπικών φορέων. Εδώ στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουμε οριμάσει και γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί αίτημα πολύχρονο. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να επιδιώξετε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις μια ερώτηση σχετικά με την κρίση των προσφύγων. Η εδαφική συνοχή δεν χρειάζεται και μια, ένα νέο προσανατολισμό όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Διότι ε, πολιτική για τους πρόσφυγες και μεταναστευτική πολιτική δεν αφορά μόνο την, ε, το επίκαιρο θέμα που είναι ένα θέμα που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, καιρό, ε, σε λίγο καιρό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένταξη, ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις μεθοριακέ περιοχές. Εκεί χρειαζόμαστε συγκεκριμένες, συγκεκριμένα μέτρα από εσά. Ευχαριστώ κύριο Έντριτ. Ευχαριστώ. Λίγο πολύ τα ίδια με απασχολούν όπως και άλλοι, αλλά από διαφορετική οπτική γωνία όπως φαντάζεστε. Για την κλιματική αλλαγή. Είσαστε πεπισμένος πόλεις σαν το Μπέρμιχαμ πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τον φόρο για την είσοδο στην πόλη, το τέλος μάλλον αυτό, στα πλαίσια των στόχων του 2020 για τους πράσινους στόχους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, η μετανάστευση. Πόσοι θα φτάσουν εδώ τελικά, μια που είναι αυξανόμενα τα νούμερα. Εσεί, πιστεύετε ότι με την καλύτερη θέληση του κόσμου, πιστεύετε ότι μπορείτε να έχετε μια περιφερειακή πολιτική και μια πολιτική συνοχή, αν δεν έχετε ιδέα για το πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν σε ποιο σημείο τη Ευρώπη, Όλη αυτή η πρότασή σα δεν έχει κανένα νόημα εφόσον δεν ξέρετε ποια θα είναι η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Κύριε Ζάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φυπουργέ που βρίσκεστε ε, εδώ μαζί μας και εκφορήσατε αυτήν την ομιλία για την πολιτική συνοχή. Και κυρίως για το γεγονός ότι θέσατε στο επίκεντρο την ε, διαστηνοριακή συνεργασία. Στην έκτη έκθεση της Κομισιόν δυστυχώς αυτό το στοιχείο έλειπε. Ωστόσο το Κοινοβούλιο στην δική του έκθεση το ξαναέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ε, το ζήτημα αυτό, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή ε, δράσεις στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής. Με τον ε, κανονισμό ETGC δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Αυτό που είπατε για παράδειγμα για τα λίματα και την διασυνοριακή τους επεξεργασία σήμερα θα μπορούσε πλέον να λυθεί αν δεν τίθενταν από εθνική πλευρά διαρκώς εμπόδια στις περιφέρειες που θα ήθελαν να συνεργαστούν. Ήμουν εισηγητής για τον κανονισμό ETDC ε και διαπίστωσα ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια ελλειπή συνεργασία μεταξύ των φορέων του Interreg και εκείνων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως νομικό εργαλείο τον κανονισμό ETGC. Ε Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να διευρυνθεί η νομική βάση για τη συνεργασία. Τέλος, το τελευταίο διάστημα βιώνουμε για άλλη μια φορά ένα κλείσιμο των συνόρων λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ωστόσο ότι η κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία για την ενίσχυση της ε, συνεργασίας των περιφερειών και τη διασυνοριακή συνεργασία. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας είναι τεράστιες. Ε, θα πρέπει να αξιοποιηθούν και γι' αυτό το λόγο αν μπορέσετε να συνεχίσετε το δρόμο που έχει ήδη χαραχθεί θα ήμασταν πολύ ευγνώμονες προς εσάς. Ευχαριστώ κύριος Ρούρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και εγώ θα ήθελα να πω στον Υφυπουργό ότι ήμουν και εγώ δήμαρχος ε, μιας μικρής πόλης και γνωρίζω τα εμπόδια και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Υπάρχουν ωστόσο και μεγάλες δυνατότητες και θα ήθελα να σας παραπέμψω και στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δήμοι και οι κοινότητες που θα πρέπει να ε, λαμβάνονται περισσότερο υπόψη για την επίτευξη των στόχων. Τώρα για τις μικρές και τις μεσαίες πόλεις υπάρχουν παραδείγματα όπου αυτό το πολυπολικό σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό αναδεικνύει και πόσο σημαντικό είναι βεβαίως ο αστικός χώρος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε την Ήπεθρο. Και εκεί υπάρχει προστιθέμενη αξία από άποψης πολιτικής εδαφικής συνοχής. Και θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω διάφο... ένα μια διαφορετική άποψη από αυτά που είπατε. Για την απλούστευση. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις, ξέρετε, ότι μερικές φορές κρατάμε το επίπεδο σφάλματος στο 2%. Αυτό σημαίνει χι εκατομμύρια για τις, από τις απάτες. Στην πραγματικότητα είναι διπλάσιο. Τι γίνεται με το θέμα της απλούστευσης και τι γίνεται με τη συγκάλυψη που υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά πολύ σύντομο, λιγότερο από ένα λεπτό. Τελευταία. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση και κύριε Υπουργέ θα ήθελα σύντομες απαντήσεις. Να προσπαθήσω. Άκουσα πολλές γερμανικές ερωτήσεις, θα απαντήσω γερμανικά. Λοιπόν, για το νέο νομοθετικό εργαλείο που χρειαζόμαστε, το συμπληρωματικό προς το ETGC, να το ξανατονίσω. Δεν θέλουμε ανταγωνιστικό εργαλείο, αλλά συμπληρωματικό εργαλείο. Στόχος μας είναι να κατασκευαστεί, να δημιουργηθεί μια δομή προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή. Χωρίς ωστόσο αυτή η νέα, αυτό τον, αυτός ο νέος μηχανισμός να δημιουργήσει νέος, νέα εμπόδια. Αν δείτε ε, αντίστοιχους μηχανισμούς που υπάρχουν στο, με έδρα το Λουξεμβούργο, μιλάμε στην ουσία για ε, δομές λογισμικού προς το παρόν. Αλλά αν δούμε τα πρώτα έργα που θα κατασκευαστούν στην πράξη ένας βιολογικός καθαρισμός για παράδειγμα ή ε, μια νέα σειροδρομική γραμμή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Λουξεμβούργο θέλει να φτιάξει ένα καινούριο τραμ. Και αυτό το τραμ θα πρέπει να περνά και τα σύνορα με τη Γαλλία. Και εκεί τα πρότυπα είναι διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το κοινοβούλιο το γαλλικό να ε, τροποποιήσει τον δικό του νόμο προκειμένου να, να υπάρξει δυνατότητα κατασκευής αυτού του έργου. Στην κυρία Μπαγασό, η γαλλική περιφέρεια που θέλει να συμμετάσχει σε ένα project τραμ κάνει ένα αίτημα στην Εθνική της Αρχή και λέει για αυτό το τραμ μέσα σε αυτή την ε, μεθοριακή περιοχή, γεωγραφικά περιορισμένη. Δεν θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε με βάση του γαλλικούς κανόνες δεν θα, ε, ή με βάση τους ε, ε, κανόνες. Δεν θα επινοήσουμε και μια τρίτη νομοθεσία που δεν υπάρχει. Θα αποφασίσουμε εάν θα ε, επιλέξουμε, θα, θα αποφασίσουμε μάλλον εάν θα βασιστούμε στη γαλλική νομοθεσία ή στη λουξεμβουργιάζικη νομοθεσία. Να πούμε δηλαδή, να πει η γαλλική αυτή περιφέρεια ότι ε, συμφωνούμε, δεν θα εφαρμόσουμε τους γαλλικούς κανόνες, αλλά τους ξεμβουργέζικους. Ελπίζω να απάντησα έστω σε έναν βαθμό στα ερωτήματά σας. Φυσικά αν έχετε τη διάθεση ε, θα μπορούσαμε να σας στείλουμε και τα σχετικά έγγραφα. Υπάρχει ένα έργο που έχουμε επιτελέσει. Ξέρουμε ότι δεν θα ολοκληρωθεί το όλο θέμα ε, στη διάρκεια της δικής μας προεδρίας γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ε, εμπόδια ακόμα. Αλλά αυτό που θέλουμε να επιδιώξουμε είναι να ε, θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανονισμός ή οδηγία που θα δίνει τη δυνατότητα στα 28 κράτη-μέλη, αν το θέλουν, να ε, ορίσουν ποια, ποια ακριβώς είναι οι τοπικοί φορείς που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ε, τα κονδύλια και τα ταμεία αυτά, σε ποιους τομείς βεβαίως, γιατί προφανώς δεν μπορεί να αφορά μια τέτοια επιδίωξη τους πάντες και όλους τους τομείς, Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι τεχνικές επιδομές, ε, υποδομές, ε, περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας, Πάρτε για παράδειγμα την εισρωή βελγικής ενέργειας, αιωλικής ενέργειας στο δίκτυο ε, ηλεκτρικού ρεύματος του Λουξεμβούργου. Πώς θα γίνει σήμερα αυτό, δεν γίνεται. Ποια, ποια θα είναι η χρέωση που θα χρησιμοποιήσουμε, η βελγική ή η λουξεμβουριανή. Για να απαντήσω και σε ένα άλλο ερώτημα δεν θα πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο μας μόνο τις διεθνείς μεταναστευτικές ροές αλλά και τις ενδοευρωπαϊκές. Και πρέπει να σας πω ότι προερχόμενος από την Ήπεθρο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίμα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο για να μετεγκατασταθούν σε πόλεις. Και Πρέπει να σας πω ότι το ίντερνετ αποτελεί την τρίτη βιομηχανική επανάσταση που μας προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες για τις μεθοριακές και τις αγροτικές περιοχές. Αν εξετάσετε προσεκτικά τις κοινωνίες μας θα δείτε ότι έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα δύο βασικές αλλαγές. Από τις κεντρικές δομές έχουμε περάσει στις αποκεντρωμένες δομές. Σκεφτείτε τι έχει γίνει στον τομέα της ενέργειας στην ε, Γερμανία εξαιρετικό παράδειγμα ε, ε, αποκέντρωσης και από τον ανταγωνισμό, η άλλη αλλαγή είναι ότι από τον ανταγωνισμό έχουμε περάσει στην συνεργασία. Δείτε και αυτήν την ε, οικονομία της κοινή χρήσης, το sharing economy, δείτε τι κάνουν οι νέοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο αλλαγές, η, η τάση προς την αποκέντρωση και η τάση προς την συνεργασία προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες στις περιοχές της υπαίθρου αλλά και για τις ε, μεθοριακές περιοχές. Πολλές φορές άλλωστε τα δύο ταυτίζονται. Πολλές ε, περιοχές υπαίθρου είναι και μεθοριακές ταυτόχρονα. Αυτό που έχω δει όμως στο παράδειγμα του Λουξεμβούργου είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αν υπάρχει ε, ε, αν οι άνθρωποι της, της οικονομίας, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι των ε, κοινοτήτων, των μεθοριακών δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν, τις ευκαιρίες που τους δίνονται, τότε δεν πρόκειται να τις αξιοποιήσουν. Ενώ αντιθέτως αν τις γνωρίζουν, τότε μπορούν να, να δημιουργηθούν και δυνατότητες ανάπτυξης. Να σας πω, η Lufthansa για ποιο λόγο έχει εταιρείε της θηγατρικές στην Ινδία. Γιατί δεν τις εγκατέστησε σε περιοχές αγροτικές ή της υπαίθρου ε, στην ε, Ευρώπη. Αυτές είναι οι μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας και όλα αυτά είναι οι εδαφικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το 2015 η πολιτική συνοχή μα δεν μπορεί να είναι ίδια με εκείνη που ήταν το 1990. Αυτό εννοώ ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική συζήτηση μακροπρόθεσμου ορίζοντα για τα σενάρια που ανοίγονται μπροστά μας. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει και σε αυτή θα επικεντρωθεί όχι μόνο η Λεξεμβουριανή ε, Προεδρία αλλά και όλο το έργο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για τι επόμενε δεκαετίε. Ευχαριστώ πολύ. Να σα ευχαριστήσω κύριε Υφυπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμβολή στην ε, συζήτησή μας. Με χαρά θα υποστηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Λουξεμβουριανή Προεδρία. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα μέλη της Επιτροπής της Περιφερειακής Ανάπτυξης με χαρά θα ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες σας. Ευχαριστούμε.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε εδώ την επόμενη προσκεκλημένη μας. Ας αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι η Επίτροπος Κρέτσου ήρθε στην συνεδρίασή μας πριν από δύο εβδομάδες για να παρουσιάσει τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιπλέον χρηματοδότηση σχέδια συνοχής στην Ελλάδα. Με την κατεπίγουσα διαδικασία. Γι' αυτό και είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση και ήρθε η Επίτροπος. Σήμερα η Επίτροπο Κρατιού έρχεται και πάλι εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία για τα 25 χρόνια του Ιντερέγ. Δημιουργήθηκε το 1990. Και τα τελευταία 25 χρόνια το Ιντερέγ έγινε ο δεύτερος στόχος της ε, πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014 με 2020 με τα διάφορα σκέλη, διασυνοριακή, διακρατική και περιφερειακή συνεργασία, στηρίζει την ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών και υπογραμμίζει ιδιαίτερα τις διασυνοριακές περιφέρειες που καλύπτουν το 7% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιντερέ καλύπτει τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις χώρες ΕΖΕΣ, την Νορβηγία, την Ελβετία και το Λίχνενστάιν, έξι χώρες ένταξης και 18 γείτονες χώρες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο προπολογισμό είναι μικρός, 3% και πιο λίγο ακόμα από το συνολικό προπολογισμό της συνοχής. Αλλά χιλιάδες προγράμματα έχουν αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών και έφτιαξαν γέφυρες ανάμεσα στους λαούς και τις ε, διάφορους οργανισμούς διαπεριφερειακά. Συνεπώς, η Επίτροπος ήρθε σήμερα για να μας μιλήσει για αυτήν την ε, πετυχημένη υπόθεση. Προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε με την παρουσίαση αυτού του success story με μία μικρή ταινία που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 You see, it, you see, it was a very short... Είδατε, ήταν μια πολύ σύντομη ταινία, αλλά παρουσιάζει μια επιτυχημένη υπόθεση. Α, σήμερα το πρωί θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Μέχρι τη μία μπορούμε να δουλέψουμε. Ακριβώς επειδή υπήρξε διακοπή κλπ πως θα δώσω το λόγο τώρα στην Επίτροπο Κρέτσου να μας παρουσιάσει αυτή την πετυχημένη ιστορία του Ιντερεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ στην Επιτροπή Ρέγγι και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη διασυνεργειακή συνεργασία που νομίζω υπό το φως των εξελίξεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Χθε ήμουνα στο Λουξεμβούργο για μια διάσκεψη ε, με την οποία γιορτάσαμε 25 χρόνια του Ιντερεκ. Εκεί συναντήθηκα με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για το Ιντερεκ και έκαναν το Ιντερεκ επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Το είδατε κι εσείς από την σύντομη ταινία ποια είναι τα επιτεύγματα θα αρχίσω την ομιλία μου σήμερα ευχαριστώντας όλους αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς. Όλους αυτούς που μέσα από το Ιντερεγ ή άλλες πρωτοβουλίες έχουν φροντίσει να έχουμε μια πιο ενωμένη Ευρώπη και να αποτελεί αυτό ένα θετικό για μας, ένα πλεονέκτημα. Όπως είπε και η κυρία Μιχαήλ πριν, το Interreg έχει αρχίσει από το 1990 και κύριος στόχος ήταν να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από την ενιαία αγορά. Για κάποιες διασυνοριακές περιοχές, στις 15 πρώτες του Interreg, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Εμείς που ερχόμαστε από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η δυναμική του Interreg είναι πιο πρόσφατη, αλλά μας βοηθάει και μας όλους να μπορέσουμε να χτίσουμε, έχοντας υπόψη μας το παρελθόν, να χτίσουμε το μέλλον για τα παιδιά μας. Το Ιντερεκ τα τελευταία 25 χρόνια έχει φροντίσει να υπάρξει τεράστια πρόοδος και αυτό έχει επιτευχθεί και με την ενθουσιώδη συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα επιτεύγματα λοιπόν αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε τώρα, γιατί τόσα πετύχαμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια τώρα να τα ξεχάσουμε. Πρώτο επίτευγμα είναι η εμπιστοσύνη. Γιατί χιλιάδες προγράμματα Interreg, πρόθεση, η ειρήνη, η συμφιλίωση, η εμπιστοσύνη είναι το βασικό για κάθε πετυχημένη συνεργασία. Και κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό που κάποιοι πιστεύουν ότι πόλεμη είναι η λύση για τα κοινά μας προβλήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κοινέ προκλήσεις ξεπερνιούνται μόνο από κοινού εφόσον σεβόμαστε την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και εφόσον είμαστε ανεκτικοί απέναντι στους πιο ευάλωτους, σε αυτούς που υποφέρουν, αλλά βέβαια προσέχοντας να υποστηρίξουμε και τη δικιά μας ε, ασφάλεια. Οι γείτονες, το είπα και χτες στο, στην Επιτροπή, ότι είναι σαν μια οικογένεια που ζούμε μαζί, γι' αυτό και πρέπει να αλληλοκαταλαβαινόμαστε και από κοινού να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Βλέπω μερικές φορές που οι χώρες δεν μπορούν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν μια κοινή πρόκληση. Και είναι θλιβερό αυτό. Το δεύτερο επίτευγμα είναι η βελτίωση της διασύνδεσης. Το Interreg έχει στηρίξει 3.500 προγράμματα από γέφυρες, ε, δρόμους κλπ. Με βελτίωση της πρόσβασης, προβασιμότητας όλων. Το τρίτο επίτευγμα είναι η υγεία. Και εδώ Έχουμε ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία ένα πολύ καλό πρόγραμμα με ένα μεγάλο και καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο. Αυτό το θέμα της διασυνοριακής υγείας είναι κάτι για το οποίο μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα στην Ουσέρδα που είναι στα Πυρηναία όπου χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση. Το τέταρτο είναι η προστασία της φύσης. Τα δάση δεν έχουν σύνορα, κινδυνεύουν από πυρκαγιές όπου και αν βρίσκονται. Είτε τα έχουν φτιάξει άνθρωποι, είτε υπάρχουν από πάντα, είτε είναι στις Άλπες, είτε είναι αλλού. Μας κάνουν να καταλάβουμε πόση δύναμη έχουμε στα χέρια μας για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Είναι σημαντικό όμως να ενώνουν τις δυνάμεις τους δεσυνοριακά οι άνθρωποι για να τα προστατεύσουν. Και το τελευταίο είναι ανάπτυξη και απασχόληση οι σχετικές πλατφόρμες που στηρίζονται με διακρατική συνεργασία δείχνουν ότι το Interreg μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά για να αντιμετωπίσει τις σημερινές μεγάλες προκλήσεις, η ανάπτυξη και απασχόληση για εκατομμύρια νέους οι οποίοι βρίσκονται χωρίς δουλειά. Χάρη στο Interreg λοιπόν πολλά προγράμματα έχουν πάρει πολιτικό βάρος. Έχουμε πάνω από 100 προγράμματα Interreg που είναι έτοιμα να επενδύσουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τους επόμενους μήνες. Γνωρίζουμε λοιπόν τα επιτεύγματα αυτά. Ξέρουμε όμως συγχρόνως ότι πρέπει να επιτευχθεί παρετέρω πρόοδος. Ξέρουμε ότι παραμένουν πολλά εμπόδια, είτε νομικής φύσεως, είτε διοικητικής φύσεως, είτε ε, προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις διασυνοριακές δραστηριότητες προτεραιότητά μου είναι να τα μελετήσω όλα και να κάνω προτάσεις. Γι' αυτό και θα υπάρξει μια διαβούλευση με το κοινό ακριβώς για τα εμπόδια που υπάρχουν στη διασυνοριακή συνεργασία. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες από την 21η Σεπτεμβρίου μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι τις 24. Θα είναι μια δημόσια διαβούλευση και όλοι θα μπορούν να απαντήσουν αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Βασίζομαι σε εσά όχι μόνο για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, αλλά για να μας προτείνετε νέες ιδέες και προκειμένου να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους που ζουν σε διασυνοριακές περιφέρειες, τους επιχειρηματίες, γενικά τον κόσμο να συμμετάσχει σε νέα προγράμματα. Θέλω και τον προβληματισμό σας λοιπόν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη διασυνοριακή συνεργασία στι περιφέρειες από τι οποίες προέρχεστε και να μας τα πείτε για να τα συζητήσουμε. Ένα άλλο θέμα είναι η μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ο κύριος Γιάφκοφτσιτς έχει την έκθεσή του για την ε, νέα στρατηγική όσον αφορά την Αδρυτική και τον Ιόνιο. Θα επανέλθω μετά. Οι μακροπεριφερειακές συνεργασίες είναι μια νέα προσέγγιση που απορρέει από την εδαφική ε, συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Αυτές οι στρατηγικές οι μακροπεριφερειακές έχουν ένα δικό τους πλαίσιο το οποίο συμφωνούν οι συμμετέχουσες χώρες και έτσι μπορούν από κοινού να έχουν μακροπρόθεσμους στόχους και να χτίσουν πάνω σε νέες ευκαιρίες. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι συμπληρώνει την παραδοσιακή εδαφική συνεργασία γιατί διευκολύνει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, στην τοπική οικονομία, ενισχύει τους ε, θεσμούς με ε, διασυνοριακή θεσμική συνεργασία και μπορεί να αποφεληθεί από διάφορες ε, πηγές χρηματοδότησης και τα κοινωνικά ταμεία, τα ζωτικά ταμεία κλπ. Ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι μάλιστα κάτι που μπορεί κάλλιστα να εμπίπτει και στο επενδυτικό ταμείο που πρότεινε ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος Γιούνκερ. Ήδη μέχρι τώρα ό,τι έχουμε είναι μια επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει την προετοιμασία και τη στήριξη των διάφορων τέτοιων μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Βαλτική και αλλού έχουμε ήδη θετικά αποτελέσματα. Η στρατηγική Αδριατική Ιουνίου που εγκρίθηκε ε, πρόσφατα είναι μια σημαντική πρόκληση. Και τέλος, η στρατηγική για τις Άλπεις εγκρίθηκε τον Ιούλιο και θα φέρει αποτελέσματα την επόμενη χρονιά. Με αυτές τις στρατηγικές μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ειδικέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ειδικέ αυτές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν χαίρεται για την σύσταση του κ. Γιάθκοφτσης που περιλαμβάνεται στην έκθεσή του όσον αφορά την Αδριατική και το Ιόνιο που έχετε σήμερα το απόγευμα. Και για αυτή τη στρατηγική αλλά και για τις άλλες στρατηγικές οι συμμετέχοντες πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν οι διοικητικοί πόροι για να τεθούν και σε εφαρμογή αποτελούν το αποτέλεσμα ετοιμάτων από τις ίδιες τις χώρες μέλη. Είναι πολύ βασικό λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις χώρες μέλη όμως για να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να ενστερνιστούν αυτές τις στρατηγικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει κεντρική σημασία ρόλο βοηθώντας τη συνειδητοποίηση και σεβόμενο τις εσωτερικές πολιτικές. Επίσης βοηθάει να προβληθούν οι στρατηγικές αυτές και τα προγράμματα και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Πιστεύουμε ότι θα γραμμιστούν έτσι καλύτερα οι εθνικές πολιτικές και τα προγράμματα προς τους στόχους των στρατηγικών. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τις υποψήφιες χώρες. Γνωρίζω ότι μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου Γιούγκερ της πολιτικής απόφασης να μην υπάρξει διεύρυνση κατά τη διάρκεια της εντολής του, όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να συνεργαστούν. Η στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, για παράδειγμα, είναι και για τις χώρες μέλη, αλλά και για μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι Υπουργοί Εξωτερικών θα καθίσουν με τους Υπουργούς Αρμόδιους για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και θα βοηθήσουν οι χώρες αυτές, οι υποψήφιες δηλαδή, να νιώσουν ότι ανήκουν και αυτές και ότι τις περιμένουμε στο μέλλον. Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή με τις στρατηγικές αυτές και είναι πολύ σημαντικό όλοι να προσπαθήσουμε να πετύχουν. Και αυτό θα γίνει βοηθώντας διοικητικά, ερμηνεύοντας και κάνοντας πράξη τις καλές ιδέες από τη θεωρία στην πράξη. Και θέλω να ολοκληρώσω αναφερόμενοι σε μια βασική ανησυχία που έχουμε αυτή την εποχή που είναι οι πρόσφυγες. Ο κύριος Γιούγκερ στην κατάσταση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι πήγε να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, ότι είναι θέμα ανθρωπιστικό, θέμα ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά ότι για την Ευρώπη είναι και θέμα ιστορική δικαιοσύνη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρο όπου όλοι μα κάποια στιγμή ήμασταν πρόσφυγε, και εγώ. Η οικογένειά μου έφυγε όταν ήρθαν οι Ρώσοι και πήγαμε στην Ρουμανία για να διατηρήσουμε τη ρουμανική μας ε, ταυτότητα. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε με τα διαστατικά και επενδυτικά ταμεία. 20 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 θα δαπανηθούν προς αυτό το σκοπό για σπίτια, για υποδομές υπέρ των ε, προσφύγων στην Ήπεθρο και στις αστικές περιοχές. Σήμερα στο Λουξεμβούργο καλώ τις διοικητικές αρχές του Ιντερέγκ για να εξετάσουμε και δυνατότητες στήριξης τέτοιων μέτρων και στα πλαίσια νέων προγραμμάτων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με την οικονομική κρίση, με την άφηξη προσφύγων, όλα αυτά ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι με συνεργασία είμαστε περισσότερο ισχυροί. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, όχι λιγότερη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Η εδαφική συνεργασία θα οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή Ευρώπη και γι' αυτό ελπίζουμε να μπορούμε να βασιστούμε στη δικιά σας τη στήριξη θα τα καταφέρουμε πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση. Thank you, Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ως συνήθως, περνάμε στις θέσεις και ερωτήσεις, καταρχήν, των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Ο κ. Βανίλ Ρόι. έχω την αίσθηση ότι εδώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Χρόνια πολλά, είδα και μια τούρτα να περνάει. Πού πήγαινε? Μια φωτογραφία τούρτας. Για τα, είναι τα κεράκια του Interreg, το, το Interreg τι μοιράζεται μαζί μας. Δεν έχουμε ένα πραγματικό κέικ. It's Έχω αυτή την αίσθηση ότι όταν εγώ εγώ την, τη δεκαετία του 90 όταν ήμουν υπουργό περιφερειών είχαμε, είχα μεγάλη πείρα από αυτό. Και αργότερα ήμουν πρόεδρος της ε, Ένωσης ε, Συνοριακών Περιοχών της Ένωσης, Διασυνοριακών Περιοχών της Ένωσης. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο πάντα έδινε έμφαση σε αυτό το τμήμα της πολιτικής συνοχής. συχνά υπήρχε αυτό και στις προτάσεις του Συμβουλίου. Υπάρχει μια σύμπνοια σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, και χαίρομαι για το μήνυμά σας. Δεύτερον, για την εδαφική συνεργασία είναι το δεύτερο θέμα. Καλό είναι αυτό που είπατε, αλλά από πίσω από αυτό που λέτε έχουμε την εδαφική συνοχή, το οποίο μας ξεφεύγει

και η οικονομική συνοχή. Το εδαφική το ξεχνάμε λιγάκι, έτσι. Τι γίνεται, τι υπάρχει από πίσω. Πώς αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Σας το λέω έτσι για να προβληματιστείτε. Τρίτον, η παρατήρησή σας για τους, ε, μετα... για τους πρόσφυγες. Γιατί επεκταθήκατε λιγάκι πέρα από το θέμα σας. Ζητάμε ευελιξία στις χώρες που έχουν προβλήματα και σε άλλες που μπορούν να αποκτήσουν. Ευελιξία. Και μάλιστα θέλουμε να μάθουμε και από την πρόταση για την Ελλάδα. Είπαμε ότι καταργείται η συγχρηματοδότηση στην περίπτωση της Ελλάδας. Η ομάδα μου, το ΕΛΚ, λέει ότι μπορούμε να βάλουμε τη συγχρηματοδότηση είναι στο 95% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Δεν κοστίζει τίποτα. Και αν η χώρα, ας πούμε, το υποστήριξει, γιατί να μην το κάνουμε. Ίσως θα πρέπει να υπάρξουν νέες προτάσεις και να καταργηθεί η χρηματοδότηση. Και κάτι, ένα θέμα επικαιρότητα. Χθε λάβαμε ε, την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την επίδοση στις δημόσιες προμήθειες. Έχουμε τέσσερις χώρες που τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Τις τέσσερις χώρες που μελετήσαμε. Μπορεί να έρθει την επόμενη φορά με ένα καλό έγγραφο που θα μιλάει για αυτό το θέμα των δημοσίων προμηθειών. Αυτό το θέμα της εξάντε ερεσιμότητας. Γιατί τότε, εάν δεν υπηρεούνται αυτοί οι όροι, θα πρέπει να σταματήσει η οικονομική ροή, τα χρήματα προς ε, την δεδομένη χώρα, προς την χώρα Χ, ας πούμε, που έχει αυτό το πρόβλημα. Όταν έχουμε συνεδριάσεις με μία επίτροπο, με έναν επίτροπο, προετοιμάζουμε πάντα την επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, Θέλω να δράξω την ευκαιρία για να σας συγχαρώ κι εγώ για τα 25 χρόνια του Interreg. Εγώ κατάγομαι από τη Σαξονία, μια περιφέρεια που συμμετέχει και μπορεί να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο Interreg ε, σε αυτήν την ε, διασυνοριακή συνεργασία και η Σαξονία για το μέγεθός της έχει, ένα πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλα σύνορα με την ε, Τσεχία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις διασυνοριακές περιοχές, μεθοριακές περιοχές. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες, τους συλλόγους, τους δήμους της κοινότητες που στην πράξη υλοποιούν αυτήν την ε, διασυνοριακή συνεργασία. υπάρχουν για παράδειγμα δίγλωση παιδικής όταν και είχαν ιδρυθεί αυτοί πριν καν υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες και πριν καν δοθούν εγγυήσει σε εκείνους που θα μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη, στις ε, ομάδες διάσωσης ανθρώπων που πολλές φορές βοηθούν ανθρώπους από την άλλη πλευρά των, των συνόρων χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει πραγματικά να ε, εργαστούμε ε, και χωρίς ή πριν μάλιστα συναυθούν και διακρατικές συμφωνίες. Και θα ήθελα να το συνδέσω και με τα θέματα που συζητήσαμε με τον εκπρόσωπο της ε, Λουξεμβουριανής Προεδρίας. Θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους επί τόπου, πολλά από τα προγράμματα δεν θα είχαν στεφτεί με επιτυχία. Και γι' αυτό απευθύνω έκκληση και προς την Κομισιόν. Ξέρω ότι έχει ήδη τεθεί στόχος να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να απογραφειοκρατικοποιηθούν ε, όσον αφορά την πρόσβαση στις, στα κονδύλια, στα ταμεία. Βρείτε τρόπους ώστε οι μικροί σύλλογοι, οι μικρές κοινότητες, οι δήμοι να έχουν τη δυνατότητα με απλοποιημένες διαδικασίες να ε, αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση χωρίς να χρειάζεται διαρκώς να περνούν από αυτές τις τεράστιες μακροχρόνιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Γιατί υπάρχουν τρόποι να ε, εξασφαλιστεί αυτό χωρίς ε, περιττή ε, γραφειοκρατία και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να πούμε και στο ελεγκτικό συνέδριο ότι το θέμα δεν είναι πάντοτε το κάθε πρόγραμμα ύψους 5.000 ευρώ να έχει αξιοποιηθεί ενδεχομένως έως το τελευταίο σέντ, το πρόβλημα, το ζητούμενο μάλλον, είναι να υπάρξουν αποτελέσματα στην πράξη. Μπορεί να γίνουν και σφάλματα, αλλά είναι ανθρώπινο αυτό. Πρέπει να μπορούν τα ταμεία, τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν στην πράξη επιτόπου στις μεθοριακές περιοχές. Για τους πρόσφυγες αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι να υπάρξουν δράσεις, πρωτοβουλίες για την καλύτερη ένταξη και ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να ενταχθούν και οι ίδιοι στη κοινωνία μας και αν υπάρχουν ε, δυνατότητες αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει ευελιξία τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μήνες, τα επόμενα χρόνια για τον σκοπό αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Χαίρομαι που θέτετε έμφαση την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη τίποτα άλλο δεν οικοδομείται. Και αυτό το λέει κάποιο που έρχεται από πρώην κομμουνιστική χώρα και καταλαβαίνει τι σημαίνει εμπιστοσύνη. Δυστυχώ σε τέτοιε χώρε ε, όλα έχουν σημασία, επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια, ε, σημασία έχει ποιο είναι στην εξουσία, ποιο κόμμα κυβερνάει και η σχέση με αυτό το κόμμα. Και μάλιστα όσοι είναι κοντά στην εξουσία εποφελούνται. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο αρμόδιος ε, στην Κομισιόν για να συλλέγει τα παράπονα των πολιτών. Γιατί συχνά ακούμε ότι δεν παίρνουν απαντήσει αυτοί οι άνθρωποι. Και όλοι θέλουν διαφάνεια. Ποιο ποιοι, με ποιον μπορούν να έρθουν σε επαφή στην Κομισιόν για να απευθύνουν τα παραπονά τους. Ο επόμενος ομιλητής. Δεν θα δώσω συνέχεια στο ερώτημα της κυρίας Τόμασιτς, γιατί εγώ ανήκω στο κυβερνών κόμμα, αλλά εγώ προσωπικά με την κυρία Τόμασιτς, ειδικά για την ε, περιφερειακή συνεργασία, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το πρόγραμμα Interreg. Γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντε, και εγώ είχα θαυμάσει εμπειρία με το Interreg. Εφαρμόσαμε 30 με 40 προγράμματα. Όταν ήμουν πρόεδρος της ε, περιοχής, της περιφέρειας Ίστρια και ασχολήθηκα προσωπικά και η συνεργασία μας με τους Σλοβαίνους και Ιταλούς εταίρους μας επέτρεψε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα και να κάνουμε ένα καλό σχεδιασμό. Σας ζητώ λοιπόν το ίντερνετ να το καταστήσετε ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες του χαρτοφυλακίου σας. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση που μπορεί να είναι καινοφανής, αλλά πέρα από τη διασυνορική συνεργασία θα έπρεπε να έχουμε και μια συνεργασία μεταξύ περιφερειών που δεν ανήκουν σε όμορες χώρες. Γιατί έχει νόημα να προωθήσουμε μια τέτοια συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, επίπεδο μεταξύ χωρών που δεν είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, που δεν είναι όμορες χώρες και που είναι χίλια, ας πούμε, χιλιόμετρα ενδεχομένως μακριά. Όμως, έχουν ενδιαφέρον για μια τέτοια συνεργασία. Πρόσφατα, άκουσα να εκφράσετε μια τέτοια επιθυμία από περιφέρειες που δεν είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεργαστούν με περιφέρειες που είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία, γιατί νομίζω ότι αξίζει να μου στηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά επίσης τη μακροπεριφερειακή συνεργασία, εδώ πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Όπως ξέρετε, το είπατε και εσείς εξάλλου, είμαι εισηγητής για τη στρατηγική Αδριατικής και Ιωνίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συντάσσοντας την έκθεση, εντόπισε τις διαφορές που έχουμε εδώ εμείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε δημιουργώντας μακροπεριφέρειες και ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό. Τι περιμένει ο κόσμος από το Κοινοβούλιο. Το κείμενο αυτό που ετοίμασα να το ψηφίσουμε σήμερα. Ετοιμάζοντάς το, άκουσα διάφορες ιδέες, τις έλαβα υπόψη μου και προτάσεις και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας αυτές για να παίρνουμε καλές αποφάσεις και για να μην, είμαστε, να μην κινούμαστε και πηγαίνουμε προς διάφορες κατευθύνσεις, γιατί αυτό συνέβη σε αυτήν την περίπτωση. Και επίσης, ε, η κρίση των ε, μεταναστών επηρεάζει πια και την Κροατία. 6.500 μετανάστες πέρασαν στην Κροατία τις τελευταίες 24 ώρες. Εμείς αρχίσαμε να υποδεχόμαστε χώρες, ε, αντίθετα από άλλε χώρε, τουλάχιστον μία χώρα που χτίζει τείχο, τείχους, τουλάχιστον η Κροατία καλωσορίζει τους μετανάστες με χαμόγελο, ετοιμάσαμε καταλήματα για αυτούς και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά όμως δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε πολύ εάν δεν μας δοθεί βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας κάνω έκκληση να μα βοηθήσετε λοιπόν, γιατί η κατάσταση θα χειροτερεύσει σίγουρα. Πολύ περισσότεροι μετανάστες θα φτάσουν στην Κροατία και μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση. Παρακαλώ, θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Όχι, συγγνώμη, ο τελευταίος συντονιστής. Κυρία Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ. Είμαστε πολύ άριθμοι εδώ οι ευρωβουλευτές που επιθυμούν ε, να ευχηθούν χρόνια πολλά στο Ίντερεγ. Όταν λέμε χρόνια πολλά σε κάποιον, καμιά φορά κάποιο, βλέπουμε ότι έχει μια θλίψη τα μάτια του. Έχω την αίσθηση ότι το ίντερνετ σήμερα είναι και αυτό θλιμμένο. Όταν βλέπουμε την ίδια στιγμή να χτίζονται τείχη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που είναι ακριβώς η αντιστροφή του πνεύματος του προγράμματος αυτού, του Interreg, που είναι να καταργηθούν τα σύνορα, να καταργηθούν τα εμπόδια, να πέσουν οι τείχοι, να υπάρξουν γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών. Επομένως, θα πρέπει να καταλάβουμε τι παίζεται σήμερα με την κρίση των προσφύγων που δοκιμάζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, λοιπόν, θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το πρόγραμμα. Που πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που είχε όραμα, που ήταν πρωτοπόρο. Όταν κοιτάμε το σύνολο των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, είπατε κι εσείς, το πρόκλημα της κλιματικής αλλαγής, τις φυσικές καταστροφές, τις προκλήσεις στον τομέα της υγείας κτλ. λοιπά Όλες αυτές οι προκλήσεις μας αναγκάζουν να δώσουμε παγκόσμιες συνολικές απαντήσεις σε κλίμακα που δεν αφορά ένα κράτος μόνο ή μία περιφέρεια, αλλά πολλές περιφέρειες και κράτη. Επόμενη παρατήρηση. Την ξέρετε, γιατί τη συζητήσαμε πλειστάκης. Είναι οι δυσκολίες που έχουν οι νησιωτικές ε, περιφέρειες και υπερπόντιες ε, περιοχές που δυσκολεύονται να υποφεληθούν 100% από τις ευκαιρίες ε, του Interreg και της διασυνοριακής συνεργασίας. Στην τελευταία διαπραγμάτευση πετύχαμε κάποια πράγματα, μια κάποια ευελιξία που μπήκε στο ίντερεγ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Τελευταίο. Συμμερίζομαι απόλυτα τη γνώμη του κυρίου Γιάκοβιτς. Δηλαδή, σήμερα Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την υποχρέωση για συνεργασία μεταξύ όμορων περιφερειών και να επιτρέψουμε μια συνεργασία μεταξύ περιφερειών που δεν έχουν κάποιο κοινό σύνορο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την έκκλησή σας για περισσότερη Ευρώπη. Πιστεύω και εγώ ότι ιδιαίτερα εδώ στο ζήτημα με τους πρόσφυγες ε, καλούμαστε να αποδείξουμε τι πρεσβεύουμε και εδώ έχει να παίξει ρόλο και η πολιτική συνοχή, όχι μόνο στο, στην ε, εδαφική ε, συνοχή αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Τώρα, για τον ρόλο της πολιτικής συνοχής θέλω να πω ότι δεν θεωρώ σωστό να χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία για μηχανισμούς κυρώσεων. Υπάρχουν στην συνθήκη τα αντίστοιχα άρθρα που προβλέπουν τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα το άρθρο 7, και η πολιτική συνοχής έχει ως στόχο την υποστήριξη των περιφερειών και όχι την επιβολή κυρώσεων σε ε, πρακτικές που δεν επιτρέπονται. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο όμως είναι αν υπάρχουν, αν υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις για μέτρα υλοποίησης και αξιοποίησης των διαστατικών ταμείων και των, του, συγκεκριμένα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την εκπόνηση μέτρων που θα έχουν ως αποδέκτες τους πρόσφυγες στις μεθοριακές περιοχές. Αυτό ε, με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ γιατί ακριβώς θα αποτελούσε την συμβολή της πολιτικής συνοχής για τη, στην αντιμετώπιση της ε, προσφυγικής κρίσης. Έχω όμως και ένα ερώτημα για το Interreg και την εδαφική συνεργασία που αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα ε, προστιθέμενης αξίας της ε, συνεργασίας σε, ευρωπαϊκής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε σχέδια για την βελτίωση ε, της ε, συνεργασίας, όχι μόνο μέσω της συνεργασίας τοπικών περιφερειών, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Και τελικό ερώτημα. Στις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο, ο προϋπολογισμός ε, για την πολιτική συνοχής περιορίστηκε. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρχουν επαρκή ε, κονδύλια στο μέλλον για το συγκεκριμένο τομέα πολιτική. Καλώ ήρθατε, Επίτροπε. Συμφωνώ με την κυρία Βάνα σε ό,τι αφορά τι ε, συμφωνίε εταιρική σχέση. Και εκεί θέλω να σταθώ λιγάκι. Οι κανονισμοί του 2014-2020 για τα επενδυτικά ταμεία λένε ότι αυτές δεν ανήκουν στις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης. Όμως οι κανονισμοί λένε ότι η συμφωνία εταιρική σχέσης θα πρέπει να δημιουργεί ε, συμπληρωματικότητα με τα προγράμματα εδαφικής ε, συνεργασίας. Η γενική σας διεύθυνση εντόπισε κάποια προβλήματα για το συντονισμό. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί ο συντονισμός. Λαμβάνοντα υπόψη ίσως και την ε, σημασία του να εμπλακούν και οι κοινωνικοί εταίροι και οι οικονομικοί εταίροι των εν λόγω περιφερειών. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλους 11 ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Ναι κύριε Μάσκουρ, σας είδα, σας έχω βάλει στον κατάλογο. Θα ήθελα να σας ζητήσω όμως να είστε σύντομοι, ένα λεπτό ο καθένας, προκειμένου να έχουμε και τον χρόνο για να μας απαντήσει η Επίτροπος στις ερωτήσεις που θα τις έχουμε θέσει. Ο κύριος Ράιμον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, δεν χρειάζεται να σας πω ότι κάποιος, ως κάποιος που έχει μεγαλώσει σε τέτοια μεθοριακή περιοχή, είμαι υποστηρικτής προγραμμάτων όπως το Ίντερικ. Θα ήθελα όμως να σας πω και εγώ, όπως και η συνάδελφος Κρέλ, ότι Πολλοί έχουν υποβάλει τα παράπονά τους σε μένα για το γεγονός ή μάλλον και την πρόθεσή τους να μην ξανασυμμετάσχουν σε προγράμματα του Ιντερεκ ακριβώς γιατί ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη από γραφειοκρατικής και διοικητικής άποψης ε, η πρόσβαση αυτή. Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι θα πω εγώ σε αυτούς τους ε, πολίτες πώς, μπορώ, πώς θα μπορέσω να τους πείσω να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα του Interreg και πώς θα τους βοηθήσουμε. Είπατε κάτι για διαβούλευση. Νομίζω ότι μια διαβούλευση δεν θα πείσει τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν ξανά στα προγράμματα Interreg. Ποια είναι συγκεκριμένα τα βήματα που θα κάνετε και που θα αναλάβετε προκειμένου να πούμε στις τοπικές κοινότητες σας παρακαλούμε συμμετάσχετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς έχει το λόγο για να υποβάλει το ερώτημά του. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα για την προσφυγική κρίση. Είμαι υπέρ. Αυτού που είπε ο συντονιστής μας. Θα πρέπει να ακολουθεί ο δρόμος που ακολουθήθηκε στην ελληνική κρίση, στην κρίση της Ελλάδας. Ήμουν και δήμαρχος στο παρελθόν και έχω εμπειρία από διασυνοριακά προγράμματα και έργα. Το πρόβλημα όμω σήμερα είναι ότι πάρα πολλά διασυνορικά έργα έχουν μείνει πίσω λόγω της προσφυγική κρίσης. Τι θα κάνετε. Για την στρατηγική, για την Αδριατική και το Ιόνιο ε, συμμετέχουν και τέσσερις ε, χώρες, ε, τρεις εκ των οποίων, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, δεν είναι ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θα συμμετάσχουν στο, στην ε, στρατηγική αυτή και η Πουγουδουμού και το Κωσυφοπαίδιο. Πώς θα διασφαλίσουμε τα κονδύλια, την επάρκεια των κονδυλίων για την ε, πολιτική συνοχή στα επόμενα χρόνια. Αυτές οι χώρες θα έχουν δικαίωμα να αξιοποιήσουν προγράμματα και κονδύλια ευρωπαϊκά. Ο κύριος Νοβάκοφ, ευχαριστώ. Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 ε, υπήρχαν, χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν 6.000 έργα ε, στον τομέα των μεταφορών. Τα περισσότερα στις φτωχές περιοχές. Ακριβώς γιατί εκεί υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί δεν έχουν τις διοικητικές δυνατότητες, τους πόρους υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σε περιοχές όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είμαστε μέλη της ε, Σέγγεν, κάτι που δυσκολεύει την κινητικότητα. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε προβλήματα με διάφορες διαδικασίες και διοικητικό άχθος που επιβάλλεται και στις δύο πλευράς των συνόρων. Γι' αυτό αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απλοποίηση. Πώς θα καταλήξουμε σε απλοποιημένες διαδικασίες εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την διασυνοριακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ε, συζήτηση, για αυτή την ε, πολύτιμη πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει και αυτό ε, τονίζεται, υπερτονίζεται και από το γεγονός ότι μόνο 30% του πληθυσμού των μεθοριακών περιοχών γνωρίζουν ότι υπάρχουν δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό είναι στην Ανατολική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση για το ίντερεκ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο αν υπάρχουν αναλύσεις για τα αποτελέσματα που έχουν αποφέρει, που έχει αποφέρει, που έχουν αποφέρει ομάδες ε, περιφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο του κανονισμού 1082 του 2006 ήταν μια πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ιντερεγ για την ενίσχυση της ε, διασυνοριακής ε, και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Γνωρίζω, ωστόσο, ότι σε πάρα πολλές... Γνωρίζω μάλιστα ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η κατάσταση έχει αλλάξει. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα απαλλαγούμε από την γραφειοκρατία. Έχω μια πρόταση. Εγώ έχω εφαρμόσει ε, προγράμματα του Ίντερεγ. Σα καλώ να δείξετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτούς που υλοποιούν τα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά... Υπάρχουν πάρα πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι τοπικοί φορείς. Αλλά όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν στις τοπικές ε, αρχές, στις εθνικές αρχές. Υπάρχουν οι έλεγκτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν τα Υπουργεία στα κράτη-μέλη. Αυτοί γνωρίζουν ποια είναι τα εμπόδια και πώς μπορούν να ε, ξεπεραστούν. Όλα αυτές οι διαδικασίες όμως απαιτούν χρόνο και έτσι οι άνθρωποι απελπίζονται. Θεωρούν ότι δεν, μπορούν, ότι δεν θα μπορέσουν τελικά να ξεπεραστούν ποτέ τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση το Interreg να λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά τα εμπόδια. Η Πρόεδρος, ε, να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να τηρείτε όλο το χρόνο για να έχουμε το χρόνο να, να ακούσουμε τις απαντήσεις της Επιτρόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, να έχουμε περιορισμένο χρόνο, θα προσπαθήσω να τον ε, τηρήσω. Μιλάμε για την 25η επέτειο γενέθλια του Ιντερεκ Ιντερεκ το οποίο έχει ενισχύσει τα διασυνοριακά προγράμματα. Μέσα σε αυτήν την μεταναστευτική κρίση εγώ θα περιοριστώ σε κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Επίτροπο. Πρώτον, τι ρόλο μπορούν να παίξουν διασυνοριακές περιφέρειες σε αυτή την κρίση. Και δεύτερον, σε τι βαθμό τα διαφορετικά ταμεία και το κοινωνικό ταμείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό, να βοηθήσουν δηλαδή στην προσφυγική κρίση. Ευχαριστούμε πολύ. Μοσκούρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Είναι ευτυχές ότι μπορούμε να γιορτάσουμε τα 25 γενέθλια του Ιντερέγκ. Εγώ σε τοπικό επίπεδο είχα κάποιες αρμοδιότητες και παρακολούθησα πολύ σημαντικά προγράμματα. Οι δύο ερωτήσεις μου είναι εξή. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι ο προπολογισμό είναι 3% μόνο από τον προπολογισμό της πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι τα έχει πάει τόσο καλά, προβλέπουμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό του Interreg. Δεύτερον, πρέπει να φροντίσουμε όλες οι δράσεις μας να έχουν σαν αποτέλεσμα περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Έχουμε πολλές δυσκολίες, οι χώρες μας δεν έχουν αρκετά οικονομικά μέσα, συνεπώς μόνο με τη βοήθεια του ίντερνετ και τα λοιπά θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τις επικράτειές μας. Ο κύριος Έκριτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ παρατήρηση θέλω να κάνω και θέλω τα σχόλιά σας από αυτής. Διαπίστωσα ότι το πρόγραμμα αυτό είναι για την κατάργηση των συνόρων στην Ευρώπη. Πολύ ωραία, εφόσον συμφωνούν οι χώρες, έχει καλώς. Αλλά αναφερθήκαμε σε νοσοκομεία διασυνοριακά. Στον Ενωμένο Βασίλειο έχουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ένα παράδειγμα με τις διαφορές του ενωμένου Βασίλειου είναι ότι ένας τεράστιος προπολογισμός και πάρα πολλοί φόροι από τους Βρετανούς πληρώνονται και πάνε στο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν υπάρχει όμως ένα τέτοιο διασυνοριακό νοσοκομείο, πώς θα πληρώνεται. Όλη αυτή η αρχή της διασυνοριακής συνεργασίας δεν καταργείται άμα είναι ένας που πληρώνει. Thank you. Thank you very much, Mr. Blanco Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χαιρετίζω τα γενέθλια αυτά, γιατί όντως τέτοια ταμεία όπως της περιφερειακής ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μετά τη συζήτηση όμως έρχομαι στην ε, διασυνοριακή συνεργασία Γαλλικίας και Πορτογαλίας. Ήταν μια από τις πρώτες τέτοιες συνεργασίες που βοήθησε την ευρωπαϊκή οικονομία και τα πράγματα επιταχύνθηκαν πολύ μέχρι να αρχίσει η οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Και όντως ε, υπήρξε πολύ καλύτερη σύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών χάρη στα προγράμματα αυτά. Τώρα, οι πόροι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν, είπαμε, και για την απασχόληση, που πρέπει να είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα. Είναι βασικό, λοιπόν, οι ευρωπεριφέρειες να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση με μια μεθοδολογία από την οποία να μπορούν να αποφελθούν όλοι. Η συνεργασία μεταξύ περιφερειών πρέπει να επεκταθεί και σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά. Να υπάρξει πιο μεγάλη μορφία στα συστήματα πληρωμών και βέβαια μεγαλύτερη κινητικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ριστία Μπόντς. Δεν πρόφερα καλά το όνομά σας μάλλον, λέει Πρόεδρος. Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Κρετού. Καλώς ήρθατε. Είπατε κάτι για γείτονε, ότι οι γειτονικέ χώρες είναι σαν τα μέλη μιας οικογένειας. Στη χώρα των Βάσκων, από όπου προέρχομαι εγώ, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε οικογένεια και γλωσσική και πολιτιστική, εθνική απ' όλα παρόλο που υπάρχουν σύνορα που χωρίζουν τη χώρα των Βάσκων με τη Γαλλία ή άλλες περιοχές. Πολλά εμπόδια υπάρχουν, τα είπατε κι εσείς, διοικητικά, νομικά. Είναι αλήθεια ότι έχουμε καλά παραδείγματα, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα και πολλά εμπόδια στην υγεία. Φαίνεται ότι λειτουργεί, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια όταν πρόκειται για την υγεία σε διασυνοριακό επίπεδο. Είπατε πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμμετοχική οικονομία σε τοπικό επίπεδο. Είναι καλό να ενισχύουν τη διασυνοριακή συνεργασία, κάτι που γίνεται και στη χώρα μου. Καλώς θα ξεκινήσει αυτή η δημόσια διαβούλευση. Εσείς μετά τι θα κάνετε με τις πληροφορίες που θα συλλέξετε από αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Εσείς τι θα προσφέρετε και τι ρόλο θα παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαχείριση των πληροφοριών που θα συλλέξετε με την διαβούλευση αυτή. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε κάθε δυνατότητα που προσφέρει η διασυνοριακή συνεργασία. Ευχαριστούμε. Τόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την κυρία Κρέτσου που ξαναήρθε μέσα σε τόσο μικρό διάστημα να μας δει. Για το Interreg θέλω να πω ότι είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το Interreg στα σύνορα Τσεχίας-Σλοβακίας και θέλω να αναφερθώ στο περιβάλλον είναι ζωτική σημασία στι διασυνοριακέ επαφέ. Η συνεργασία μεταξύ περιφερειών μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά, αλλά μόλις υπάρχει ένα πρόβλημα στον αέρα από εκπομπές ή ρήπανση ποταμών ή μετά από πλημμύρε, όλα αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν το περιβάλλον και συχνά ζημιώνουν τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο να σκεφτεί μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη συνεργασία. Τέλος. Από πλευρά αλληλεγγύης απογοητεύτηκα από την ψηφοφορία γιατί ήμουνα μόνο ένας από τους τρεις που στήριξε την πρόταση της Επιτροπής. Δρέπομαι γιατί η πολιτική συνοχής σημαίνει άρση εμποδίων και ενίσχυση της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση, κυρία Μαλέτσου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κυρία Επιτρόπε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που συχνά αναρωτιέμαι και εγώ για την εδαφική συνεργασία. Πώς μπορεί να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη και πώς μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και θα σας δώσω το παράδειγμα της Κροατίας για την περιφερειακή αυτή συνεργασία. Το Interreg είναι ένα πρόγραμμα μέσα σε άλλα προγράμματα για την δαφική συνεργασία και στην Κροατία έχουμε τέσσερα διασυνοριακά διεθνικά αλλά και διαπεριφερειακά σύνορα. Ήξερα για το τελευταίο τι είναι το Ιντερέκ και Turbo. Όταν όμως μιλάμε με τους τελικούς δικαιούχους, αποθαρρύνονται αμέσω. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα, τόσε πολλέ κατευθυντήρε γραμμέ, τόσα πολλά σημεία αναφορά που αλλάζουν που δεν παρακολουθούν πια. Ίσως χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και η προσέγγιση να είναι τέτοια που να καταλήγει σε κάτι ενιαίο και να μην κατακαιρματίζεται. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τις απόψεις σας. Τώρα, 10-12 λεπτά μας μένουν για να μας απαντήσει η Επίτροπος. Σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η σημερινή μας συνάντηση και θα προσπαθήσω να σας πω και εγώ κάποια σχόλια στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πάντως όλους για τα θέματα που θέσατε, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια. Για την ε, εδαφική συνοχή, συμφωνώ, δεν ταυτίζεται με την εδαφική συνεργασία και ελπίζω στην 7η πολιτική συνοχή, σε αυτή η, δια... η διάσταση της εδαφικής συνεργασίας να συμπεριλαμβάνεται. Σχετικά με την ευελιξία, τέθηκε ως θέμα από πάρα πολλούς συναδέλφους. Όπως είπα και στην ομιλία μου, η αντιμετώπιση το... της μετανάστευσης είναι σημαντική και χρειάζεται αυτή τη στιγμή να εξασφαλιστεί ε, αυτό που προβλέπουν και οι κανονισμοί, η επαρκής ε, ευελιξία, αλλά αφορά και τα κράτη-μέλη τα ίδια. Αν δείτε την Ιταλία και την ε, Ελλάδα, στην Ιταλία έχουν αξιοποιηθεί τα ταμεία, ενώ στην Ελλάδα καθόλου. Εμείς επικεντρώνουμε την, στην ένταξη. Δεν ε, στοχεύουμε σε συγκεκριμένη μειονότητα. Στόχος των ταμείων, των κονδυλίων αυτών είναι να βοηθηθούν ε, μειονεκτούσες περιφέρειες και περιοχές όπου ζουν και μετανάστες. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ταμεία, το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο περιφερικής ε, ανάπτυξης προκειμένου να προχωρήσουν πολιτικές ένταξης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αν όμως θεωρούν ότι χρειάζεται τροποποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων, τότε τα κράτη-μέλη μπορούν να το κάνουν. Έχουν τη δυνατότητα αυτή. Κρίνεται κατά περίπτωση. Όπως γνωρίζετε, εμείς συγγραμματοδοτούμε προτεραιότητε και όχι συγκεκριμένα έργα. Γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν ε, επιστροφή χρημάτων για μεταναστευτικά προγράμματα στο 100%. Αυτό που χρειάζεται να διασφαλίσουν εκείνα είναι ότι θα ε, συμπεριλαμβάνουν τα προγράμματα αυτά επιλέξιμες ε, δράσεις. Εμείς προσφέρουμε και καθοδήγηση και στήριξη προ τα κράτη-μέλη, ενημερώνουμε τι ακριβώ μπορούμε εμεί να χρηματοδοτήσουμε και τι όχι. Και ήρθα εδώ σήμερα για να σα πω μεταξύ άλλων ότι αντιμετωπίζουμε και χειριζόμαστε τα αιτήματα τροποποίηση πάρα πολύ γρήγορα όταν υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη. Γνωρίζω ε, ότι η έκθεση ε, του Ελληνικού Συνεδρίου υπευλήθη και δημοσιεύτηκε χθε και Θα τα συζητήσουμε αυτά και το Δεκέμβριο. Πάντως, Κομισιόν και Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν τον ίδιο στόχο. Την ε, εξασφάλιση της ε, εφαρμογής της ε, πολιτικής συνοχής μέσω του προϋπολογισμού. Και βεβαίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο συνολική συζήτηση ε, και στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κυρία Κρέλ, να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα τώρα. Η κυρία Κρέλ έχει δίκιο. Οι τροποποίησεις που γίνονται στις ζωές των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους είναι μεγάλες εξαιτίας του Ιντερεκ είναι κάτι που πρέπει να το συζητάμε περισσότερο. Εγώ προσπαθώ να πηγαίνω σε όσο γίνεται περισσότερες χώρες και να βλέπω τα προγράμματα επιτόπου. Πήγα λοιπόν και, στην, ε, και στα σύνορα τα γαλλογερμανικά, αλλά και αλλού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου και την ιστορία, γιατί μιλάμε εδώ πέρα γιατί μιλήσαμε μάλλον πριν για την Κροατία, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα γαλλογερμανικά σύνορα βέβαια τώρα είναι σε ειρήνη και είναι πάρα πολύ ωραία πως οι άνθρωποι περνάνε από, το ένα, από μια πλευρά στην άλλη χωρίς πρόβλημα. Το ίδιο ανάμεσα στην Πολωνία και τη Γερμανία όπου πάνε και επισκέφτονται φίλους από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι καθημερινά. Όσον αφορά τώρα την απλοποίηση, ναι, οι δημοτικές αρχές συνεργάζονται και πρέπει να συνεργάζονται. Η... Το διοικητικό άχθος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές συνεργάζονται. Οι χώρες πρέπει επίσης να κάνουν μια προσπάθεια απλοποίησης. Πρέπει να αντισταθούν στην ε, τάση που υπάρχει να προσθέτουν επιπλέον εθνικούς κανόνες. Η απλοποίηση είναι μεγάλη ευκαιρία και ελπίζω ότι για τη νέα προγραμματική περίοδο θα έχουμε νέους κανόνες πιο απλούς. ήδη από του χρόνου. Η... Το είπε και η κυρία Τόμασίτς, το είπα και εγώ ότι η εμπιστοσύνη είναι ζωτική σημασία. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για τούρτα γενεθλίων, πρέπει να ξέρουμε ότι φτάνουμε εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλιώς δεν θα γινότανε. Τώρα με ρωτήσατε πολλά πράγματα όσον αφορά το ρόλο των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πράγματι, οι οργανώσεις της κοινωνίας των ε, πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχει και διαβούλευση. Εμείς πάντως στη γενική μας διεύθυνση τι θέλουμε αυτή την προσέγγιση και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές γιατί πιστεύουμε ότι παίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Εγκρίθηκαν ακριβώς επειδή χώρες μέλη το ζήτησαν. Συνεπώς, οι χώρες μέλη πρέπει να φροντίσουν για την απλοποίηση ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν πρόσκοπτα. Όσον αφορά τώρα την Κροατία πιο συγκεκριμένα, ναι, είναι μια νέα κατάσταση, ένα νέο παράδειγμα για τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και χαιρετίζω τον τρόπο, τον πολιτισμένο τρόπο με τον οποίο η Κροατία υποδέχεται τους πρόσφυγες που ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι ο κανόνας αν δεν θέλουμε οι προσπάθειες που κάναμε τα 25 αυτά χρόνια να πάνε χαμένες. Οι προκλήσεις όντως δεν έχουν σύνορα. Ούτε ο αέρας, ούτε το κυκλοφοριακό, ούτε θεομηνίες, τίποτα. Οι άκρος περιφερειακές περιοχές είναι αλήθεια ότι είναι μέσα στην περίμετρο του Interreg. Πάντα μπορούμε να κάνουμε βέβαια ακόμα καλύτερα. Πάντως, ναι, οι άκρος περιφερειακές περιοχές είναι μέρος των προγραμμάτων μας και τις μεταχειριζόμαστε επίσης όρους. Για να απαντήσω τώρα στο σχόλιο της κυρίας Βανά, συμφωνώ μαζί της. Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής είναι ξεκάθαρος οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, μείωση των διαφορών μεταξύ των περιφοριών και δεν θέλουμε βέβαια η συνοχή να στραφεί σε βάρος των χωρών μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αντίθετα, πρέπει να τις βοηθήσουμε μέσω της συνοχής, ιδίως τις χώρες που βρέθηκαν σε μια εκτακτή κατάσταση. Η απειλή απόσυρση των διευθυντικών ταμείων δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ούτε και νομικά στέκει, ούτε και πολιτικά πιστεύω. Συνεπώ. θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ψύχρεμα την κατάσταση. Όσον αφορά τώρα το σχόλιο της κυρίας Αμάτο, ο συντονισμός, ναι, είναι σημαντικός. Η κοινωνία των πολιτών είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και όπως έλεγα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν στις επιτροπές επιλογής για τα προγράμματα 2014-2020. Όπως έχω πει εγώ προσωπικά και εκ μέρους των περιφερειών, αγωνιζόμαστε γι' αυτό καθημερινά. Περιμένουμε πολλά από τη δημόσια διαβούλευση. Μερικές φορές ε, λυπάμαι που δεν μιλάμε συχνά για την συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Ταμείων στη ζωή των ανθρώπων. Στην Ελλάδα πήγα και μίλησα με έναν δημοσιογράφο και του έλεγα πώς έχει αλλάξει η Ελλάδα από τότε που έγινε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μίλησε, το στο παράδειγμα του μετρό της Αθήνας. Και μου είπε, ναι, ναι, το έχω ακούσει ότι έχει συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το 95% της χρηματοδότησης του μετρό της Αθήνας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψή σας για το ότι είναι σημαντικό ότι σε αυτήν τη δημόσια διαβούλευση πρέπει να συμμετέχουν όλοι όλοι όσοι δουλεύουν γνωρίζουν τα θέματα αυτά. Έρχομαι τώρα στην διακρατική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και τρίτων χωρών. Εδώ πρόκειται για τη στρατηγική Αδριατικής και Ιωνίου. Όσον αφορά αυτή τη στρατηγική λοιπόν υπάρχουν οι πόροι. Υπάρχουν πόροι και από τα περιφερειακά, αλλά για τα Δυτικά Βαλκάνια πρόκειται για τις σχέσεις καλής γειτονίας. Είναι ένα ειδικό κονδύλι. Κάποιος αναφέρθηκε στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Πράγματι, πρόκειται για περιφέρειες που έχουν ε, χαμηλότερη διοικητική ικανότητα, περιορισμένη από άλλες. Και ακριβώς γι' αυτό πιστεύω ότι η διοικητική ικανότητα είναι βασικό. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, το λέω ότι είναι μάλιστα κάτι πιο σημαντικό και από τα χρήματα. Τα χρήματα δεν είναι το παν. Υπάρχουν παραδείγματα χωρών που πήραν χρήματα αλλά που δεν μπορούν να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά, τα οποία μένουν μπλοκαρισμένα στις τράπεζες εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί δεν έχουν τη διοικητική ικανότητα να τα απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Άρα η διοικητική ικανότητα των χωρών αυτών πρέπει να βελτιωθεί. Τώρα, μερικά πράγματα που επανέρχονται. Ο κύριο Μασκάδο αναφέρθηκε στον προπολογισμό. Ο προπολογισμό εγκρίθηκε. Αλλά μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν τον προπολογισμό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για μας στην Επιτροπή το σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τα αποτελέσματα από τα κονδύλια αυτά. Και ήθελα να αναφερθώ και στα σύνορα μεταξύ της Αιχίας και Σλοβακίας, γιατί μου μιλήσατε για αυτό το παράδειγμα ε, τα προβλήματα που Και είναι παντού. Εμείς συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Βέλα προκειμένου να βρούμε κοινέ λύσεις βασιζόμενες στην αλληλεγγύη. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Είναι σαφές, είναι προφανές ότι κάποια εμπόδια ε, δεν μπορούν ε, να εξαφανιστούν ποτέ. Για παράδειγμα το γλωσσικό. Αλλά τα 25 αυτά χρόνια έχουμε κάνει τεράστια βήματα. έχουν αλλάξει νοτροπίες στις διασυνοριακές περιφέρειες. Οι ρυθμίσεις εκατέρωθεν των συνόρων έχουν ευθυγραμμιστεί. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει εκπονηθεί. Μερικές φορές βέβαια παραμένουν προβλήματα είτε διοικητικά είτε άλλα στις διασυνοριακές περιφέρειες. Η συζήτηση όμως που κάνουμε είναι σημαντική και η επέτειος αυτή των 25 ετών δείχνει ότι μπορούμε πάντα να έχουμε την κατάλληλη λύση για κοινέ προκλήσεις. Θα πάω στη Βιέννη σύντομα για τα 25 χρόνια διασυνοριακής συνεργασίας. Όλα τα λειτουργικά προγράμματα σχεδόν εγκρίθηκαν φέτος που είχαν να κάνουν με τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Ελλάδα, Σερβία για παράδειγμα, Αλβανία, Βουλγαρία. Πρέπει να δώσουμε παραπάνω σημασία σε αυτά, γιατί υπάρχουν περιφέρειες που έχουν γίνει πιο σημαντικές εξαιτίας της επικαιρότητας. Και εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε την εμπειρία. Αλλά και επί τόπου μπορείτε να αποτελέσετε πηγή πλούτου. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία Επιτροπής Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου όλων των συναδέλφων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και μπορούμε να προετοιμάσουμε βεβαίως και την επόμενη μας συνάντηση. Είστε ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε. Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες στις 3 το απόγευμα. Φέρτε τις κάρτες σας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Κυρίσω λοιπόν τη λήξη της πρωινής μας συνεδρίασης.